Εγώ, εγώ.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 μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας σήμερα και σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στον κυβερνόχωρο και σε web streaming μέσω του, της, του ιστόχωρου του Κοινοβουλίου. Πρώτο σημείο ημερήσια διάταξη, αν έχετε αντίρρηση, εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 2 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου Εάν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνεδρίασης δεν υποβληθεί καμία ένσταση, δεν έχετε αγγλικά. Τρίτο σημείο της ημέρας διάταξης είναι οι ανακοινώσει μου. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει ένσταση, θεωρούνται εκτιμένα τα πρακτικά. Αν δεν υπάρξει ένσταση μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, όπω είπαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα αλβιονικά τα οποία δεν ακούγονται. A ver, bueno. Ya, a ver si ya funciona. Sí. Λειτουργούν τώρα, εντάξει. Τρίτο σημείο της μέσης διάταξη είναι η ανακοινώση τη προεδρία. Και θέλω να σα ανακοινώσω ότι σήμερα έχουμε ένα κοκτέιλ το οποίο κανονικά προσφέρεται από το Προεδρείο για το τέλος του έτους θα είναι στην αίθουσα 4 του εστιατορίου των βουλευτών στις 6.30. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι και φυσικά και οι διερμηνείς. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4. Η νέα όθηση στη στρατηγική για την αηφόρα ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής δικτυοκαλλιέργειας με εισηγητή τον κύριο Μιλάνα. Έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις για το θέμα αυτό στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας, όχι πάντα με αρκετό χρόνο και είχαμε υποσχεθεί να είναι σήμερα το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη η έκθεση του κυρίου Μιλάνα. Νομίζω ότι όλοι έχετε διαβάσει το έγγραφο εργασία του, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλε τι γλώσσε και χωρί περαιτέρω χρονοτριβή δίνω το λόγο στον κύριο Μιλάνα για να μα παρουσιάσει το έγγραφό του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το συζήτησαμε ήδη δύο φορές το κείμενο αυτό. Σήμερα η πρόθεσή μου είναι να μην το ξανασυζητήσουμε τρίτη φορά, αλλά να δούμε τι θα βγει από τη συζήτηση που θα γίνει. Σύντομα θα σας περιγράψω το έγγραφο, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο να ακουστούν τα σχόλια των συναδέλφων. Είναι ένα πρώτο έγγραφο εργασίας. Πρέπει να αλλάξει, γιατί συνεχώς προστίθενται νέα στοιχεία στο φάκελο, ξεκινώντας από τα γενικά. Η βασική επιλογή του εγγράφου αυτού, μετά από τις δύο συζητήσεις, συναντήσεις, είναι να οριστούν οι όροι έτσι ώστε στον τομέα αυτό να υπάρξει ένας κανονισμός. Όχι γιατί η Ένωση θέλει να νομοθετήσει, γιατί η δατοκαλλιέργεια καλύπτει από τους κανονισμούς. Αυτά τα λέει το έγγραφο στις πρώτες σελίδες. Και θα προσθεθούν και επιπλέον στοιχεία στο τελικό έγγραφο σχετικά με αυτό. Δηλαδή σε άλλες οδηγίες υπάρχουν μικροσημεία ή και μεγάλα σημεία που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια. Η ανάγκη για κανονισμό έγκυται στο να δημιουργηθούν οι νομικοί όροι που από τη μία μεριά θα εναρμονίζουν τα εργαλεία που υπάρχουν στην νομική αγορά της Ένωσης, ας το πω έτσι, και από την άλλη να έχουμε την επικοινωνία, δηλαδή να καλυφθεί ένα χάσμα που υπάρχει στην ανάπτυξη αυτού του οικονομικού τομέα. Η ανάπτυξη αυτή τα τελευταία χρόνια σημείωσε αύξηση και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα τα νομικά εργαλεία δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί στην Ένωση ο τομέας αυτός με τους ίδιους ρυθμούς. Θέλουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να καλύψουμε την καθυστέρηση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. όσον αφορά την αύξηση της παραγωγής, που να καλύπτει μια αντικειμενική έλλειψη στην Ένωση, μια έλλειψη περίπου 1.300.000 τόνους και κατανάλωση που ξεπερνάει τους 500.000 τόνους. και θα έχουμε και επιπλέον αύξηση της αγοράς από τον ΦΑΟ, ΕΕΦΣΕ και λοιπά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δηλαδή μας λένε ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση της αγοράς του προϊόντος της υδατοκαλλιέργειας. Και υπάρχει και μία μείωση των αποθεμάτων των ψαριών ανοιχτής θάλασσας. Άρα, η επιλογή εκ μέρους της Ένωσης πρέπει να είναι στρατηγική. Γι' αυτό το κείμενο πρώτον καταγράφει την κατάσταση, δεύτερο περιγράφει την νομική και οικονομική κατάσταση του κλάδου αυτού και τρίτο επισημαίνει τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν όσον αφορά τις προοπτικές. Και λέμε ότι ο κανονισμός είναι το εργαλείο μέσω του οποίου μπορούμε να περάσουμε στη νέα αυτή φάση. Σας είπα ήδη ότι η ανάπτυξη, του τομέα στην Ένωση αυτή ήταν μικρή. Το 2002 και τα διάφορα εργαλεία που είχαμε από τότε μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν έτσι ώστε στην Ένωση να έχουμε μια τάση αυξητική του τομέα αυτού αντίστοιχο με τη ζήτηση. Αυτό θέλουμε, να είναι αντίστοιχη με τη ζήτηση. Άλλο βασικό θέμα, γιατί το πρώτο ήταν αυτό, η ενεπαρκής αύξηση ανάπτυξη. Θα δούμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. η υδατοκαλλιέργεια επιδέχεται πολύ υψηλές επενδύσεις και υπάρχει και ισχυρή τεχνολογική διάσταση. Μία εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας στοιχίζει πολύ και η απόδοσή του μέσω μακροπρόθεσμη. Και ίσως γι' αυτό δεν είχαμε αυτού του είδους την ανάπτυξη, διότι δεν υπήρξε ένα σημαντικό δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίως είχαμε μερικές μεγάλες μονάδες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα είδους συγχρηματοδότηση ή να γίνει πιο ευέλικτη τέλο πάντων η χρηματοδότηση και οι επενδύσει. Έπειτα η δεδοκαλλιέργεια δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν τα υδατοκαλλιέργεια των ψαριών της θάλασσας, των γλυκών νερών, των μαλακόστρακων. Δηλαδή μέσα στην υδατοκαλλιέργεια των ψαριών της θάλασσας υπάρχουν πολλές οικογένειες ψαριών με διαφορετικές τεχνολογικές απαντήσεις και διαφορετικές οικονομικές απαντήσεις ως προς τον κύκλο του προϊόντος και ως προς τις αγορές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή να μιλάμε για το Σολομό ή για άλλου είδους ψάρια, πέστροφες κλπ. έπειτα υπάρχουν σοβαρά διοικητικά εμπόδια. Υπάρχουν δηλαδή άκαμπτοι κανόνες, μερικές φορές εκ μέρους Ένωσης, ή καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα. Τίποτα ουσιαστικά δηλαδή δεν επιταχύνει την επιχειρηματική δράση. Και δεν μιλάμε για την αγορά, μιλάμε για τα διοικητικά εμπόδια που πολλές φορές με την βραδύτητα που δημιουργούν αποτρέπουν τις επενδύσεις. Έπειτα έχουμε ένα, θα το έλεγα, αστικό έλλειμμα. Δηλαδή ούτε στα κράτη, στις περιφέρειες, στις επιμέρους κοινότητες δεν υπάρχουν στοιχεία που να εξασφαλίζουν τους όρους ώστε να ξέρουμε πού να γίνει, πού να τοποθετηθεί η νέα μονάδα, γιατί και μια μικρή μονάδα ιδιωτοκαλλιέργειας έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Γιατί υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας του πέριξ περιβάλλοντος. Υπάρχουν ή όχι ρεύματα. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ρήπανση. Αυτό ξεπερνάει δηλαδή του υδατοκαλλιέργεια. Μπορεί να έχει επιπτώσει στον τουρισμό, στην ε, καλή ποιότητα των ακτών και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Μετά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την τυπολογία του προϊόντος. Έχουμε άμεσο ανταγωνισμό σήμερα σε κάθε μορφή είτε εξαγωγών είτε εισαγωγών προς την Ένωση. Από προϊόντα που προέρχονται από χώρες οι οποίοι είχαν πολύ ψηλότερους δείκτες ανάπτυξης από ό,τι εμείς, όπως η από Ανατολή, Βιετναμ, Κίνα δηλαδή, αλλά και η Τουρκία και η Χιλή, που αυτές τις τεράστιες επενδύσεις που έκαναν, και οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής, βρήκαν εύκολη είσοδο στην αγορά μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Πέρα από αυτά που ξέρουμε όλοι, δηλαδή μεγαλύτερο κόστος εργατικά, μεγαλύτερο κόστος στο ότι είμαστε βιομηχανοποιημένοι δύση, ό,τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει κόστος παραγωγής και εργατικά για μας. Έχουμε λοιπόν έναν ανταγωνισμό που πολλές φορές επηρεάζει και την ασφάλεια. Δηλαδή, έχουμε κανονισμούς που περιορίζουν την είσοδο προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο ορισμός όμως αυτών των προδιαγραφών έχει όρια. Έπειτα, η έλεγχη στα χιλιάδες σημεία εισόδου αυτών των προϊόντων δεν είναι έλεγχη καλού επίπεδου. Έχουμε λοιπόν ορισμένους εμείς περιορισμούς ή όρια όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων, το περιβάλλον, τη σχέση μεταξύ της ποσότητας που παράγεται και της ποσότητας την, την ένταση, ας το πούμε, της παραγωγής, ποσότητας νερού κλπ. Όλα αυτά είναι εκτός ελέγχου. Οπότε η καλή ποιότητα του προϊόντος μας πρέπει να κινηθεί με βάση πρωτοβουλίες που θα κάνουν το προϊόν πιο ανταγωνιστικό ή τουλάχιστον αναγνωρίσιμο. Το συζητήσαμε αυτό. Έχουμε την πολιτική ποιότητας, αλλά έχουμε και τα εμπορικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε το ευρωπαϊκό σήμα στην παραγωγή μας. Και στο έγγραφο έχω βάλει και αυτά τα δύο στοιχεία. Και το σήμα για την βιομηχανική υδατοκαλλιέργεια και για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια το σήμα. Έτσι ώστε την προστιθέμενη αξία που έχουμε με βάση την τεχνολογία μας τον έλεγχο του κύκλου παραγωγής να φροντίσουμε όλα αυτά τα μέτρα ο καταναλωτής να τα ερμηνεύσει ως προστιθέμενη αξία σε σχέση με το εισαγόμενο προϊόν. Χρειάζεται μια πολιτική σήματο που βέβαια δεν γίνεται με τρει σειρέ ένα κείμενο. Χρειάζεται εμβάθυνση. Και μετά χρειάζεται η εφαρμογή του κανονισμού. Άλλο θέμα, ευαίσθητο και λεπτό, είναι η ευζοία των ζώων μέσα στον κύκλο παραγωγής. Βέβαια γι' αυτό είναι συνυπεύθυνοι πολλοί άλλοι παράγοντες, οδηγίες ας το πούμε. Καμία όμως από μόνη της δεν ορίζει ένα πλαίσιο του, των ψαριών για τα οποία συζητάμε. Των ειδών μάλλον για τα οποία συζητάμε. Παράδειγμα, πριν από μερικές εβδομάδες συνάντησα μια ένωση φιλοζώων Άγγλων που μου είπανε και αυτό απλώς το υπενήσουμε σε ένα σημείο, μου είπαν «Ναι, πρέπει να δείτε και το πώς το προϊόν της υδατοκαλλιέργειας πώς θανατώνεται. Παρέμεινα έκπληκτος. Ένα ψάρι πεθαίνει, βγαίνει από το νερό και πεθαίνει. Όπως όλα τα ψάρια. Δεν ξέρω να υπάρχει άλλο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ξέρω. Μου είπανε, μου εξήγησαν ότι υπάρχει ένα σύστημα θανάσης. Άμεση ψήξη που κάνει τον θάνατο λιγότερο δυνηρό. Γιατί όταν βγαίνει το ψάρι από το νερό, πνίγεται. Αν το ρίξει όμω αμέσω σε μείον 8 βαθμούς πεθαίνει αμέσως και δεν υποφέρει πολύ. Στην Ευρώπη μας λοιπόν υπάρχουν και τέτοιου είδους ευαισθησίες. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ορίσουμε, να νομοθετήσουμε ακόμα και γι' αυτό. Δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε. Να έχουμε το λιγότερο ανηλές, ανηλεή τρόπο θανάτωσης των ψαριών. Συνήθω ο κόσμος θεωρεί ότι το ψάρι πεθαίνει επειδή το ψάριψε κάποιο. Ωστόσο, υπάρχει αυτό το θέμα της ευζοία των ζώων, που θα πρέπει να οριστεί με παραμέτρους που θα υπάρχουν στον κανονισμό. Επειδή έχουμε και το, τη φάση που το ψάρι είναι ακόμα ζωντανό. Η πυκνότητα των ψαριών, παραδείγματο χάνει σε μια καλλιέργεια. Να είναι πιο σωστή. Βέβαια θα λέγει κανείς δεν είναι όλο το ίδιο, δεν μπορεί να οριστεί το πόσα λίτρα χρειάζεται ένας σολομός ή ένα άλλο είδους ε, ψάρι ας πούμε, μερλούκιος κλπ. Μπορούν όμως να οριστούν παράμετροι, όχι αυστηροί κανόνες, αλλά γενικές παράμετροι που να σχετίζονται, να συνδέονται με την τυπολογία του εκτρεφόμενου είδους. Όπως με την κτηνοτροφία ξηράς, που δεν εφαρμόζει το ίδιο παραδείγματο χάρη για το αρνί ή για το μοσχάρι. Και τα δύο είναι θηλαστικά και τα δύο έχουν τέσσερα πόδια και τα δύο τα τρώμε τελικά αλλά η εκτροφή του καθενός είναι διαφορετική. το καλλιέργειο το ίδιο. Θεωρείται ένα είδος κτηνοτροφίας της θαλάσσης, ας το πούμε. Μόλις τις ιδιομορφίες της. Το να μιλάμε για την ευζοία των ζώων και των ψαριών στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ επιφανειακό. Επιφανειακό όμως δεν είναι. Θα έλεγα μάλιστα η ευζοία αυτή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Δηλαδή είναι ένα είδος ανθρωπιστικής δράσης και έναντι των ψαριών, αλλά έχει και οικονομική αξία, γιατί περνάει στην αξία του τελικού προϊόντος. Ένας εμπειρογνώμων μου εξήγησε ότι όταν τρώμε ένα ψάρι στο εστιατόριο, αν η ραχοκοκαλιά του ψαριού είναι λίγο στραβή, αυτό σημαίνει ότι εξετράφει σε, ένα, σε μια δετοκαλλιέργεια εσφαλμένου τύπου. Δηλαδή είχε πολύ λίγο χώρο το ψάρι αυτό και αναγκάστηκε να υποστεί λόρδος ή τέλο πάντων κάτι στρέβλωση της πονδυλικής του στήλη λόγω της πίεσης. Πολλά μου εξήγησαν οι εμπειρογνώμονες. Αν δω ψάρι με στραβή κοκοκαλιά, να το μυρίσω και τότε θα διαπιστώσω ότι το ψάρι αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι τόσο καλό όσο ένα που έχει την ραχοκοκαλιά ευθεία. Δηλαδή και τα οργανοληπτικά και τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά ενός ψαριού που μογάλωσε σε στενό χώρο φαίνεται. Δηλαδή και η ραχοκοκαλιά του είναι στραβή, αλλά και το ψάρι δεν είναι καλό. Άρα η ευζοία του ψαριού, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι υπερβολικό ως απέτηση έχει σχέση με μια συγκεκριμένη οικονομική αξία όσον αφορά το τελικό προϊόν. Μίλησε για τις εισαγωγές. Σε άλλη έκθεση θα συζητήσουμε νομίζω για το επίπεδο των εισαγωγών. Οπότε περνάω στο επόμενο θέμα. Μερικές συγκεκριμένες προτάσεις. για το γενικό πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο έχει στόχο την εναρμόνιση αυτών που ισχύουν, απλοποίηση των ε, διαδικασιών και όρια που θα επιτρέψουν να περάσουμε σε μεγαλύτερη και καλύτερη ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόρους. Δηλαδή, να μπούμε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως λειτουργήσαμε στην πρώτη δεκαετία, ορίζοντας κανόνες και παραμέτρους και προδιαγραφές, αλλά χωρίς να επενδύσουμε πόρους και κονδύλια, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι στη δεύτερη αυτή δεκαετία. Πενιχρά. Θα πρέπει όλα αυτά να συνοδεύονται από κονδύλια. Γι' αυτό αναφέρω την ανάγκη για ένα ταμείο, ειδικό ταμείο. Σε αυτή τη φάση δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Είναι κάπως πρόωρο. Έπειτα θα είναι ένα νέο ταμείο που ξέρετε θα σα κάνει να σα σηκωθούν οι τρίχε, Να φτιάσουμε ένα νέο ταμείο για την υδατοκαλλιέργεια που αναφέρεται τελείω ε, μη πραγματοποιήσιμο. Ή θα μπορούσε να είναι κάτι ειδικό μέσα στα πλαίσια του Ταμείου Αλίας. Πάντως ανάγκη υπάρχει. Αν θέλουμε να δώσουμε μια όθηση στον τομέα, όπως μας λέει η ανακοίνωση της Κομισιόν, μας ζητάει δηλαδή να φροντίσουμε να δοθεί αυτή η όθηση. Ε, λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει μια οικονομική υποστήριξη. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις γνώμες της Προέδρου, των Συμπροέδρων, των Επιτρόπων, δηλαδή να οριστεί αυτός ο πόρος. Αυτή η ανάγκη υπάρχει τώρα. Το αν θα είναι ταμείο αν θα είναι ένα επιμέρους ταμείο σε ένα, στα πλαίσιο που ήδη υπάρχει κάτι άλλο, αυτό το συζητάμε. Η καλλιέργεια. είναι και μια ευκαιρία ανάκτησης δράσης όσον αφορά την κλασική αλία που μειώνεται λόγω της συνολικής πολιτικής αλίας ανάκτηση όσον αφορά την ε, εργασία. Δηλαδή, αλλοίς που δεν βρίσκουν απασχόληση τοπικά μπορούν εντό εισαγωγικών να γίνουν υδατοκαλλιεργητέ. Οπότε μπαίνει το θέμα κατάρτιση. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ταμεία και μορφές υποστήριξης της κατάρτισης αλλά στο κοινωνικό ταμείο. Μια συγκεκριμένη πολιτική κατάρτισης που θα έχει σαν στόχο να αναγνωριστεί ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα του αλλιέα σε σχέση με το ιδιωτοκαλλιεργητή. Με πολύ ψηλότερη τεχνολογία. Είναι διαφορετικό φυσικά και από την χερσαία εκτενοτροφία. Δηλαδή ένα επαγγελματικό προφίλ συγκεκριμένο που να συνοδεύεται και από αντίστοιχη κατάρτιση. Πρέπει να έχουμε μία δικλίδα ως λύση ατόμων που φεύγουν από την κλασική γεωργία για οικονομικούς λόγους και που θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό το νέο πλαίσιο του ιδετοκαλλιεργητή χωροταξικό σχεδιασμός. Μόνο το σεβισμό για τις αρμοδιότητες που έχουν οι περιφέρειες κλπ. Γιατί η υποκορικότητα υπάρχει σε κάθε τομέα, σε οποιαδήποτε επιλογή και αν κάνουμε. Αλλά ο σχεδιασμός, ο χοροταξικός είναι κλειδί προκειμένου να κατευθυνθούν σωστά οι επενδύσεις. Βλέποντας τι ισχύει σήμερα, διαπιστώνω ότι υπάρχει και ανάπτυξη να αναπτυχθούν μικρομεσαίες μονάδες στις ακτές και άλλες μονάδες offshore, δηλαδή στη θάλασσα. Επιβάλλεται λοιπόν η ανάγκη όλα αυτά να είναι συμβατά, γι' αυτό χρειάζεται σχεδιασμός. Να υπάρξουν λοιπόν οι πολιτικές ώστε να την ποιότητα, όπου το σύνολο όλων αυτών των δράσεων, σύν το σήμα το οποίο ανάφερα, Έπειτα έχει, υπάρχει το θέμα της ε, τεχνολογικής καινοτομίας. ως μια συνιστόσα που θα επιτρέψει μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας που να ανταποκρίνεται σε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή στην καλή μεταχείριση των ζώων, ε, στο σωστή διατροφή κλπ. Και αυτό θα ορίζει το πώς θα χρησιμοποιείται αυτό το ταμείο. Όχι ταμείο που να μοιράζει λεφτά, να παρακολουθεί την εφαρμογή των συγκεκριμένων στόχων. Κατάρτιση. Σχεδιασμός. Τεχνολογική καινοτομία. Έπειτα ο έλεγχος ποιότητας των εισαγωγών. Σήμερα γίνεται μόνο ποσοτικός έλεγχος. Ποιοτικός έλεγχος δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν εργαλεία που να μας επιτρέπουν από τη στιγμή που έχουμε ορίσει τα πρότυπά μας μέσα στην Ένωση, να φροντίζουμε έτσι ώστε το προϊόν που εισάγεται, ανάλογα με τον τύπο που έχει, να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Και τέλος υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι δολοφόνοι της θάλασσας, τα ηχθιόφάγα, πτηνά, ουσιαστικά οι Κορμοράνη Είναι πρόβλημα αυτό. για την σημερινή δεδοκαλλιέργεια. Μεγάλη ζημιά. Και εδώ χρειάζεται σχεδιασμός για τους κορμοράνους. Υπάρχει νομίζω ένας κανονισμός. Έχουμε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Το τελευταίο, τελευταίο. το θέμα της διατροφής. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Το ψάρι τρώει ψάρι. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινή σκέψη που λέει επειδή τα ψάρια τρώνε ψάρια, τι εξυπηρετεί να ψαρεύουμε το ψάρι για να το δώσουμε να το φάει ένα ψάρι σε ιδετοκαλλιέργεια. Λάθος. Λένε εγώ νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες με βάση τις οποίες οι ζωικές πρωτεΐνες που χρειάζονται για να ζήσει το ψάρι μπορεί να υπάρχουν και φυτικές πρωτεΐνες που να υποκαταστήσουν τις ζωικές. Δηλαδή, καλλιέργειες φυτικές που θα μας δίνουν φυτικές πρωτεΐνες που μπορούν να μετατραπούν σε ηχθιάλευρα ηχθιοτροφές. Και αυτό έχει σχέση, μάλλον τίθεται εδώ το θέμα της ποιότητας των ε, ηχθιοτροφών. Πολλές φορές η εθνική νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη το προϊόν διατροφής των εκτρεφόμενων ζώων. Ε, ξέρουμε τι έγινε με τις τρελές αγελάδες όσον αφορά τη διατροφή τους. Βέβαια, αυτά δεν πρέπει να τα ζούμε ως περιορισμό, γιατί κάτι που εκτρέφεται σε μερικά χιλιόμετρα από εδώ, δεν ξέρουμε τι τρώει και δεν ξέρουμε τελικά τι μπαίνει στη δική μας τροφική αλυσίδα. Γι' αυτό θα ήθελα και γι' αυτό το θέμα και η Κομισιόν και η Επιτροπή μας σήμερα να το σκεφτεί αυτό σοβαρά και σε καμία περίπτωση να μην λειτουργήσει ως φρένο. Σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ Πάντως ε, μίλησα λιγότερο από ό,τι στις δύο προηγούμενες συναντήσεις μας. Σας καλώ όλους με βάση αυτό το σχέδιο κειμένου να μου στείλετε τις επόμενες εβδομάδες γιατί έχουμε ακόμα μερικούς μήνες καιρό να είστε γενναιόδοροι απέναντί μου με προτάσεις. Αλλά ταυτόχρονα την υπόψη την ευαισθησία ορισμένων σημείων. Χρειάζεται δηλαδή να δείξουμε ένα πνεύμα διαλλακτικό όλοι μας προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή δυνατόν θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μιλάνα. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα έχετε τον χρόνο στον απαραίτητο και νομίζω ότι τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι αυξημένες αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, φέρνουν μαζί τους και μεγάλες υποχρεώσεις και ευθύνες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι συζητούμε σήμερα για ένα τομέα όπως η υδατοκαλλιέργεια ένα τομέα ο οποίος δεν έχει τύχει της πρέπουσας προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προσπαθεί να βρει το ζωτικό του χώρο μεταξύ αλληλείας, γεωργίας, οικολογίας, τουρισμού, ανταγωνισμού από τρίτες χώρες κτλ. και ο οποίος παρόλα αυτά τα πηγαίνει σχετικά καλά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δυστυχώς μια στασιμότητα στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καν αυτάρκης αφού τα δύο τρίτα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προέρχονται από τρίτες χώρες με αλλιεύματα αμφίβολης ποιότητας που συχνά παράγονται χωρίς σεβασμό στους περιβαντολογικές υποχρεώσεις ή τους κανόνες ευημερία και υγιεινής που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Επιτροπή Αλίας η υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Έχουμε την ευκαιρία να επαναθεμελιώσουμε τον κλάδο ώστε να αποτελέσει ένα πρότυπο βιώσιμη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το επιχειρήσουμε. Άλλωστε, είναι σαφές ότι η δατοκαλλιέργεια άπτεται πολλών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας, της προστασίας των καταναλωτών, Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και που μπορεί να αποτελέσει μια ικανοποιητική αναλλακτική απάντηση στα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελία. Καλωσορίζω λοιπόν το έγγραφο εργασία του συναδέλφου κυρίου Μιλάνα, ο οποίος μέσα σε ένα σύντομο κείμενο κατάφερε να παρουσιάσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αλλά και να οριοθετήσει άξονες δράσης. Θετικά βλέπουμε την προοπτική θέσπιση ενός κανονισμού. Κάτι τέτοιο δεν αντίθετο στην αποκεντρωμένη προσέγγιση που προωθεί η αναθεωρημένη κοινή αλλιευτική πολιτική. Θεωρούμε ότι μέσα από μια κοινή ευρωπαϊκή θεώρηση του τομέα, ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας θα μπορέσει να αναβαθμιστεί. Σκεπτικοί είμαστε για την ίδρυση Ενό Ταμείου Προστήριξης της υδατοκαλλιέργεια. έχω την εντύπωση ότι με περαιτέρω συζήτηση θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ακριβώς ποιο είναι το μοντέλο που ο κύριος Μιλάνα μας εισηγείται. Τέλος, θα σχολιάσω την ευαισθησία που επέδειξε ο εισηγητή για τον τρόπο θανάτωση των ψαριών. Είμαι βέβαιος ότι σε ένα μελλοντικό κόσμο, δεν ξέρω ύστερα από πόσα χρόνια, οι άνθρωποι, οι μελλοντικοί άνθρωποι θα πληροφορούνται ότι σήμερα τρώμε έμβιους οργανισμούς για να τραφούμε και θα του σηκώνεται η τρίχα όπως ακριβώς μας σηκώνεται η τρίχα σήμερα στην ιδέα του κανιβαλισμού. Υπ' αυτή την έννοια οποιασδήποτε πράξεις ανθρωπισμού σε αυτή την πρώιμη βάρβαρη ανθρώπινη κατάχρηση άλλων βιολογικών ειδών είναι καλοδεχούμενη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιλάνα για μια πληρέστατη και καλή έκθεση. Ήταν καιρός να κάνουμε μια τέτοια έκθεση. Το γεγονός ότι ήδη στις πρώτες φράσεις της έκθεσης εξηγεί ο εισηγητής πώς αφήσαμε την υδατοκαλλιέργειά μας να λιμνάσει μεταξύ του 2001 και του 2008, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος προχώρησε με γοργά βήματα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της συζήτησης. Έχουμε μία ακτογραμμή στην Ευρώπη που είναι ιδανική για υδατοκαλλιέργεια. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να αναπτύξουμε σε ιδανικές συνθήκες την υδατοκαλλιέργεια και την ηχθειοκαλλιέργεια. Αφήσαμε όμω χώρε όπω η Χιλή, η Κίνα, το Βιετνάμ να πάρουν το πάνω χέρι σε ό,τι αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια σε παγκοσμίο επίπεδο. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τον Ρίτσι Φλίν, ο οποίο εκπροσωπούσε του Ιρλανδού ηχθειοκαλλιεργητέ σε μια ακρόαση ενώπιον τη επιτροπή μα, να μα λέει ότι ο λόγο για αυτή την εξέλιξη είναι το γεγονό ότι προτού να μπορεί ένα καλλιεργητή στην Ευρώπη να πουλήσει έστω και ένα ψαράκι έχει να ικανοποιήσει 400 κανονισμούς από τρεις γενικές διευθύνσεις, περιβάλλον, εμπόριο, θαλάσσια θέματα. Η γραφειοκρατία λοιπόν τους πνίγει κυριολεκτικά. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι είναι ιδανική ευκαιρία με αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, γραφειοκρατία και να έχουμε μια ενιαία θηρίδα για τους ε, υδατοκαλλιεργητές ώστε να μην βρίσκονται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Μιλάνα, νομίζω πολύ σωστά είπατε ότι οι αυστηροί κανονισμοί τους οποίους εφαρμόζουμε στα δικά μας προϊόντα ηχθειοκαλλιέργειες πολλές φορές δεν αφορούν τα εισαγόμενα προϊόντα υδατοκαλλιέργειες και όπως ελέγχθη, δύο τρίτα από τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εισάγουμε. Είχαμε μια πρόσφατη σύντομη συζήτηση, οπότε τέθη το θέμα του παγκασίου από το Βιετνάμ. 60.000 τόνου αυτού του ψαριού εμείς ε, εισαγάγαμε από το Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έρχεται από τεράστια τεράστιες εγκαταστάσεις βιομηχανικές στον ποταμό Μεκόγκ, ο οποίος είναι ο πιο ρυπασμένος ποταμός στον κόσμο. Είναι ένα είδος ψαριού, ένα, μια μορφή παγάσιου στο Βιετνάμ, που περιλαμβάνει, όπως έχουμε δει από τις αναλύσεις, διοξίνες, ε, ε μη αποδομούμενα πλαστικά κτλ και ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι αλείς κάνουν ενέσεις στα ψάρια από αποξηραμένα γυναικεία και μόνο ούρα για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους σε αυγά και ώστε να μπορέσει ο γόνος ο οποίος προέρχεται από αυτά τα αυγά να αναπτυχθεί ταχύτερα. Αυτά τα ψάρια λοιπόν εισάγονται στην Ευρώπη όταν εμείς δένουμε χεροπόδαρα τους δικούς μας ηχθειοκαλλιεργητές με χιλιάδες κανονισμούς. Αυτό είναι ένα έσχος. Θυμάμαι στην εποχή που ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας όταν μου έλεγε η Κομισιόν ότι το βοδινό κρέας από τη Βραζιλία εκπληρούσε όλες τις προδιαγραφές για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι στέλνανε πάντα επιθεωρητές στη Βραζιλία για να ελέγξουν την ποιότητα αυτού του βοηού κρέατο και μετά είδαμε ότι μάλλον το αντίθετο συνέβαινε και το βοδινό από τη Βασιλεία ήταν ιδιαίτερα ύποπτο και παρήγετο σε επικίνδυνες συνθήκες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Κομισιόν πράττει τα απαραίτητα για να επιθεωρήσει τις ιδιοκαλλιέργειε Παγκασίου στο Δέλτα του Μεκόγκ, που είναι η κύρια πηγή τροφοδοσίας στην Ευρώπη. Αυτό ουσιαστικά υπονομεύει την αγορά μας. Ε, δεν εμποδίζει στους, ε, εμποδίζει στους να αγοράζουν καθαρά ψάρια από την αλία ή από τις δικές μας ηχθειοκαλλιέργειες. Πρέπει λοιπόν να τονίσω ότι υποστηρίζω απόλυτα τους αυστηρούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα, όπως είπε και ο κύριος Μιλάνα. Θέλουμε τα ψάρια μας να εκπληρούν τις πιο υψηλές δυνατές προδιαγραφές, αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τους κανονισμούς μας, ώστε να μην κάνουμε τη ζωή των ε, αλίων μας, των ε, ηχθειοκαλλιεργητών αδύνατη και να του θέτουμε σε μειονεκτική θέση με την αναγωνιστικότητα. Τώρα το θέμα τη πυκνότητα και του τρόπου φώνευση των, ψάριων, των ψαριών. Αν υπάρχει πολύ μεγάλη ε, πυκνότητα σε μία δεξαμενή, η παραγωγή μειών στους σολομούς δεν είναι στο κατάλληλο επίπεδο και καταλήγει κανείς σε ένα σπογγόδες ε, κρέας αυτών των ψαριών που δεν είναι ευχάριστο στον καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η κατάλληλη ε, πυκνότητα ώστε τα ψάρια να μπορούν να κολυμπούν και να αναπτύσσουν το μυϊκό του σύστημα. Για του τρόπου φώνευση, το να βγάζουμε τα ψάρια από το νερό και να τα αφήνουμε να πεθάνουν από ασφυξία δεν είναι ο καλύτερο τρόπο, Υπάρχουν πολλέ μέθοδοι φώνευση. Η αναισθητοποίηση χρησιμοποιείται πολύ συχνά και η ΕΦΣΑ, η Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έχει κάνει μια έρευνα μεθόδων θανάτωσης για οκτώ από τα πιο συνηθισμένα θαλάσσια είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ βρίσκω προβλήματα με όλες αυτές τις μεθόδους θανάτωσης και έχω ζητήσει να υπάρξει βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η θανάτωση αυτών των ψαριών. Θέλω λοιπόν να ενθαρρύνω τον κύριο Μιλάνα να εξετάσει λίγο περισσότερο τα θέματα αυτά και να εξασφαλίσει καλύτερη θανάτωση και περισσότερη ευσοία των ψαριών. Σε ό,τι αφορά την ε, εκτροφή αυτών των ε, ψαριών. Υπήρξε μεγάλη βελτίωση γιατί υπάρχουν τώρα πολύ φυτικά, πολλά φυτικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ενώ στο παρελθόν ήταν ηχθιάλευρα και ηχθιέλαιος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% στο παρελθόν στην εκτροφή των ε, ψαριών. Έχει μειωθεί τώρα αυτό στα 50%, αυξάνει το ποσοστό φυτικών πρωτεϊνών, αλλά δεν μπορείτε να έχετε χόρτο φάγα ψάρια. Ένα ψάρι πρέπει να είναι ψαρένιο. Μπορούμε να βελτιώσουμε ίσως το ποσοστό των φυτικών προϊόντων στα ψάρια, αλλά τα ψάρια χρειάζεται να έχουν πρωτεΐνες από ψάρια στην ε, εκτροφή τους. Σε ό,τι ε, αφορά τις ε, εισαγωγές από το Περού και από άλλες χώρες, όταν εμείς θέλουμε να απαγορεύσουμε την απόρριψη ψαριών βάσει της κοινής πολιτικής, Έχουμε ένα εκατομμύριο τόνους απόρριψης ψαριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιτρέψουμε στους ε, αλείς να συλλέγουν αυτά τα προϊόντα, αυτά τα ψάρια, τα οποία είναι εκτός ποσοστώσεων ή είναι πολύ μικρά, μπορούμε στη συνέχεια να τα χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ηχθιαλεύρων και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε στη συνέχεια να εκθρέψουμε τα ψάρια στα ε, ιχθυοκαλλιέργειε και όχι απλώς να πετάμε τα ψάρια αυτά τα οποία είναι ήδη ψόφια και να μολύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται λοιπόν οι επεξεργασίες, τα υπολείμματα των ψαριών που τρώμε, όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να διατρέφονται τα ψάρια σε υδατοκαλλιέργειες. Είναι ένας τρόπος λοιπόν ο οποίος είναι πάρα πολύ ασφαλής για την εκτροφή των ψαριών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία. Θα σας παρακαλούσα να είμαστε πιο σύντομοι γιατί έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Σάντσες Περσέδο Λεβίν, Πατραονέβες, Τεσπαρέα και εγώ ο ίδιος. Εγώ ίδια. Σάντσες Περσέδο και παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όντω να είμαι σύντομο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μιλάνε για το έγγραφο εργασία που μα παρουσίασε. Υπάρχουν τρία τμήματα διαφορετικά, με διαφορετικούς προβληματισμούς και προτάσεις. Η υδατοκαλλιέργεια βέβαια έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην επικαιρότητα σήμερα είναι η αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων που μας έρχονται από τη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα τον ανταγωνισμό με προϊόντα που μας έρχονται από τρίτες χώρες. Χρειάζεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Νομίζω ότι τρεις ε, δρόμους έχουμε. Το ένα είναι η ανάπτυξη. Χρειάζεται φυσικά νομικό πλαίσιο, οικονομική στήριξη και μέσα. Πολύ σημαντικό όμως είναι να έχουμε και τη συμμετοχή του κλάδου. Δεύτερος δρόμος που πρέπει να δούμε είναι η ισορροπία με άλλες πολιτικές. Πολιτικές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την υγεία ή άλλες δραστηριότητες. Πώς θα συμβιβάσουμε δηλαδή τη γεωργία με άλλες δραστηριότητες ώστε να μην έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε ανταγωνισμό με αυτήν συνέχεια. Και τέλος, θέλουμε ανταγωνιστική γεωργία. Έχουμε ποσοστώσεις πολύ περιορισμένες, αν τις δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης πρέπει να επιμείνουμε πολύ στην ποιότητα. Ποιότητα και των υδάτων, αλλά και των τροφίμων, αλλά και των μεθόδων που έχουμε για την υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει λοιπόν να βαθύνουμε περισσότερο σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και το τελευταίο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η ενημέρωση του καταναλωτή, γιατί όλα αυτά για να πάρουν την αξία που τους πρέπει πρέπει να αξιολογούνται βάσει κάποιων δικτών. Να υπάρχει κάποια σήμανση έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει για το κάθε προϊόν από πού έρχεται, σε ποια νερά έχει καλλιεργηθεί, με ποια διαδικασία κλπ. κλπ. Είναι ζωτική σημασία και αυτό το θέμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ε, κύριε Λεβά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιλάνα, σα ευχαριστώ για την έκθεση αυτή που τη βρήκα πράγματι πολύ σημαντική. Το άγγραφό σα εγώ το βρίσκω εξαίρετο πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ καλή ιδέα να προτείνουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και να έχουμε ένα σύστημα σήμανση που να προστατεύει το περιβάλλον όσον αφορά τα ψάρια που μα έρχονται απ' έξω. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδεικνύουμε ότι εμεί παράγουμε την αλία μας με έναν πιο οικολογικό τρόπο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάντως, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε, όπως μας προτείνετε κι εσείς, να επιμείνουμε στην έρευνα πιο πολύ. Να δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη νέων ειδών, να δούμε επίσης τι γίνεται με την προστασία των ζώων, την υγεία των ζώων. Όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει το πρόβλημα να δούμε πώς θα παράγουμε τα τρόφιμα, τις ε, τροφές από τις οποίες ε, θα τρέφονται τα λιεύματά μας. Χαίρομαι πάντως που βλέπω ότι επιμένετε πολύ για το θέμα αυτό της τροφής. Να υπογραμμίσω όμως και κάτι. Το θέμα της επάρκειας, κατά πόσο υπάρχει επάρκεια στην Ευρώπη δυσκολευόμαστε τα τελευταία 15 χρόνια να διαχειριστούμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε μείωση κατά 20% της παραγωγής στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει αύξηση του στόλου. Αν μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και για την υδατοκαλλιέργεια. Σίγουρα υπάρχουν όρια. Πόσο δηλαδή μπορούμε να λιεύσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε και στην υδατοκαλλιέργεια ψάρια. Στη Βαλτική θάλασσα, στη Σουηδία πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει σε αυτό το τομέα. 60% ε, των ηχθείων πολιεύονται, προορίζονται για την υδατοκαλλιέργεια. Να ξέρετε ότι επίσης χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή ε, τροφής για τα ψάρια. χάνουμε πάρα πολύ. Μη διαχειριζόμενη καλά την κατάσταση και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έπειτα για το πρόβλημα των ασθενειών και της ευημερία των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να βρεθεί μια λύση. Πρόσφατα πήγα στην Ορβηγία, επισκέφθηκα εκεί καλλιέργειες Σολομού και διαπίστωσε ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική εκεί από ότι εδώ. Εκεί διαφοροποιούνται πάρα πολύ τα είδη. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε να μην υποφέρει το ψάρι, να λάβουμε υπόψη μας και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που έχουν να κάνουμε αυτό. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εκατομμύρια για την υδατοκαλλιέργεια. Εδώ το 2003 ανακαλύψαμε μία νέα ασθένεια στο γάδο και διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές μπορεί πολύ γρήγορα να μεταδοθεί. Στην Νορβηγία αναγκαστήκανε να σκοτώσουν πάρα πολλά ψάρια για να αποφύγουν την μετάδοση αυτή της νόσου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα προλαμβάνουμε αν θέλουμε να αναπτύξουμε καλά την εδατοκαλλιέργεια. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς των ε, ψαριών. Γιατί ορισμένα μπορεί να στρεσάρονται πάρα πολύ κατά τη μεταφορά μέχρι να πάνε στο σημείο που θα θανατωθούν. Και σίγουρα υπάρχει και μεγάλη θνησιμότητα. Και επηρεάζει το στρες αυτό τη γεύση του ψαριού. Όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα χειριζόμαστε τα ψάρια αυτά. Αν θέλουμε περισσότερα, πρέπει να φροντίσουμε να συλλέξουμε και περισσότερες γνώσεις. Πάντως ένα ψάρι να ξέρουμε ότι μπορεί να υποφέρει εξίσου όπως και ένα τετράποδο. Το έχουν αποδείξει αυτό επιστημονικές ε, μελέτες. Αν το δεχτούμε λοιπόν αυτό το στοιχείο, θα πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε με τα ψάρια αυτά που αλλιεύονται από την υδατοκαλλιέργεια σε σύγκριση με αυτά που αλλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα. Τέλος, Εδώ μιλήσαμε και για κάποια πουλιά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να χειριστούμε στην έκθεσή σας. Πάντως πρέπει όντω να υπάρχει ένα σχέδιο για να προστατεύονται και αυτέ οι περιοχέ περιοχές υδατοκαλλιέργειας. Είναι πολλοί οι οποίοι πρέπει να λάβουν το λόγο, πολλοί βουλευτέ, Κομισιόν και φυσικά ο συγητή. Σα παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Κυρία Παντράου Νέβη. <clears throat> Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη όσο το δυνατό, λέει η κυρία ναι. Πατράου Νέβε. <clears throat> Φυσικά θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντα τον κύριο Μιλάνα για την εργασία του. Μου φαίνεται ότι πάρα πολύ αξιέπαινη, πάρα πολύ κατανοήσιμη και σαφής και που δίνει την πρέπουσα έμφαση στα βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό της υδατοκαλλιέργειας. Εξάλλου, όπως είπε, είπαν και πολλοί ομιλητές, δύο τρίτα των ε, ηχθείων που καταναλώνουμε τα εισάγουμε. Επομένως, το μέλλον είναι η ιδεατοκαλλιέργεια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θέλουμε να το κάνουμε αυτό, βάσει ποιων κανόνων, με ποια μορφή θα γίνει αυτή η ανάπτυξη. Αυτό ακριβώ είναι το διακυβευόμενο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, εξάλλου σε μεγάλο βαθμό εγώ <clears throat> προσυπογράφω αυτά που ακούσαμε. Θέλω να είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία, μια μεγάλη συνένεση για την προβληματική που περιστρέφεται γύρω από την έκθεση του κ. Μιλάνα και εγώ προσωπικά συμφωνώ με τα, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ε, έκθεσης, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω μια άλλη πτυχή του θέματος που μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική. Θα περιοριστώ λοιπόν σε αυτό. Για το θέμα των εισαγωγών, ξέρω ότι αναφέρθηκε αυτό ήδη, αλλά δεν είναι περιττό να τονίσω επιπλέον ότι όταν εμείς εισάγουμε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που υπόκεινται σε διαφορετικούς φυτοϊγειονομικούς κανόνες, κανόνες ευζοίας, κανόνες περιβάλλοντος και επομένως έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, το αποτέλεσμα είναι ότι όλα αυτά έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Και ενδεχομένως αυτός είναι ο λόγος, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί Ευρωπαίοι ε, αλληλείς βλέπουν την υδατοκαλλιέργεια σαν μια απειλή για την επιβίωση του αλληλευτικού τομέα. Πάρα πολλοί λοιπόν έχουν μια αρνητική στάση σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια. Αλλά τόνισε ο κύριος Μιλάνα ότι στην πραγματικότητα η υδατοκαλλιέργεια και αναφέραμε και την υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια μπορεί να είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτούς τους ε, ε οι οποίοι έχουν όλο και μικρότερα αλλιεύματα από την κανονική διαδικασία της αλίας. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να κατανοήσουν οι αλλοίς ότι η δατοκαλλιέργεια είναι συμπληρωματική με την αλία και ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητας των αλιών και όχι μονάχα μια απειλή. Φυσικά χρειάζεται μια διαδικασία πιστοποίησης, χρειάζεται να υπάρχει ένα σύνορο κανόνων και ο κύριος ε, Στίβενσον τόνισε τη σημασία του να ξέρουμε πού αλλιεύονται τα ψάρια σε τι συνθήκες και τέλος, μια τελευταία παρατήρηση που έχει να κάνει με το ότι είναι απαραίτητο να επιμείνουμε έναντι των κράτων μελών να αντιμετωπίσουμε με ταχύ τρόπο την, τον εντοπισμό των περιοχών που είναι οι πιο πρόσφερες για την υδατοκαλλιέργεια και έχουν το λιγότερο κίνδυνο αρνητικής αλληλεπίδρασης με άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν εκεί η χώρα. Σε ένα από τα εργαστήρια τα οποία οργανώθηκαν στον τομέα της αλίας υπήρχαν παρόντες εκπρόσωποι από τη Μαδέρα, από τα, τις Κανάριες νήσους, τις Αζόρες και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τον τρόπο με τον οποίο τα Κανάρια νησιά μέσα σε λίγα χρόνια αύξησαν εκθετικά την παραγωγή τους στον αγροτικό τομέα, στον ιχθυοκαλλιεργητικό ε, τομέα μάλλον και η Μαδέρα ενώ έχει μείνει πίσω προχωράει με γόρκα βήματα Τώρα, στις Αζόρες βρισκόμαστε ουσιαστικά στο μηδέν σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι τεράστια η αποκλειστική οικονομική ζώνη των Αζωρών. Μία τελευταία λοιπόν τώρα πάλι παρατήρηση που θέλω να αναφέρω και δεν είναι περιττό αυτό το οποίο θα σας πω είναι η ανάγκη να υπάρξει και επιστημονική έρευνα για να υποστηριχθεί η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας. Τονίστηκε από την αρχή ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρέπει να κινηθούμε προς την υδατοκαλλιέργεια. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η κίνηση, αυτή η έρευνα θα πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα. Όπως είπα, το να υπάρξει μια χαρτογράφηση των περιοχών οι οποίες είναι πιο πρόσφορες για την υδατοκαλλιέργεια, αλλά συγχρόνως να υπάρξει και μια έρευνα της τροφικής αλυσίδας για τα προϊόντα αυτά, όταν μιλάμε για τα ηχθιάλευρα, είναι απαραίτητο να δούμε σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητο να έχουμε συνθετικές τροφές σε εργαστήρια, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να έχουμε μια εναλλακτική διατροφή για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και πρέπει επίσης να δούμε ποια άλλα θαλάσσια είδη μπορούν να εκτραφούν σε συνθήκες ε, υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τα χορτοφάγα θαλάσσια είδη και να έχουμε είδη τα οποία έχουν ένα δίκτυο μετατροπής πρωτεϊνών που να είναι πιο χαμηλός από αυτόν που έχουμε σήμερα και φυσικά είναι λαθασμένο να θεωρεί κανείς ότι είναι απαραίτητο να τρών τα ψάρια ψάρια και υπάρχει πάντα η δυνατότητα τα ψάρια, τα ηχθιάλευρα να αναμειγνύονται με άλλες ζωικές τροφές. Εξάλλου δεν είναι μόνο τα ψάρια τα οποία τρώνε ε, ηχθιάλευρα και πολλά άλλα ζώα τα οποία τρέφονται με ηχθιάλευρα. Θέλω λοιπόν μετά από όλα αυτά και πάλι να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή, ο οποίο μα επιτρέπει να δούμε με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στον τομέα τη υδατοκαλλιέργεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Άντρε Παρέα, σα παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ναι, θα είμαι σύντομη. Λοιπόν, η Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ε, έχει κάνει πολύ σημαντική έκθεση γιατί θα το πρέπει να αποτελέσει μέρος της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γιατί, γιατί είναι πολύ σημαντική πηγή διατροφής του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Προσφέρει εγγύσει στον κόσμο. Έπειτα βοηθάει στην ανάπτυξη. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να συμβιβάσουμε την αλλία με το περιβάλλον. Το περιβάλλον ε, μας ενδιαφέρει, Πρέπει να το προστατεύσουμε και να φροντίσουμε να κάνουμε αξιολόγηση περιβάλλοντος για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να αποτελέσει η αλία μέρος της κοινή αλευτικής πολιτικής. Η δατοκαλλιέργεια δηλαδή να αποτελέσει μέρος της ΚΑΠ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω επίση να συγχαρώ τον κύριο Μιλάνα. Ήταν πολύ καλά διαρθρωμένη η έκθεσή του και ήταν ευανάγνωστη και περιλαμβάνει πάρα πολύ θετικές πληροφορίες. Η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας πολύ καλός τρόπος να έχουμε φτηνά και υγιή ψάρια και νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια εναλλακτική λύση με την τωρινή μορφή των, της αλίας. Ήδη ο σύντροφος Στίβενσον τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη πληροφόρηση και διαφώτιση του καταναλωτή. Αναφέρομαι στο παράδειγμα το οποίο, το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ σε αυτό, αλλά είναι απαραίτητο να μην εμποδίσουμε την υδατοκαλλιέργεια με ιδιαίτερα αυστηρού κανονισμού, αλλά παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να έχουμε λογικού κανόνε. Για μένα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η κατάρτιση των ατόμων τα οποία ασκούν την υδατοκαλλιέργεια να υπάρξει ένα συγκεκριμένο προφίλ εκπαίδευσης για τα άτομα αυτά και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν και άτομα με υψηλά προσόντα τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν <clears throat> αυτή την επαγγελματική προβληματική της υδατοκαλλιέργειας. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να μπορέσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθορίσουμε ένα προφίλ κατάρτισης για τους υδατοκαλλιεργητές. Επίσης είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια σωστή χωροταξική αντιμετώπιση, να υπάρξει ένα είδος θαλάσσιας χωροταξίας για τις περιοχές όπου θα μπορέσει να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια με έναν τρόπο που θα είναι τακτικός και οργανωμένος. Και αυτό φυσικά απαιτεί μια παρακολούθηση και σε επιστημονικό επίπεδο και εγώ θεωρώ ότι είναι επίσης απαραίτητο να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες προστασίας της υγείας και της ευζοίας των ψαριών. Κύριε Μίλαν και, Μιλάνα και εγώ θέλω να κάνω μερικά σχόλια. Ήδη στο ειδικό ταμείο που έχετε ζητήσει εσείς για την υδατοκαλλιέργεια. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό ούτε καν αν είναι απαραίτητο. Γιατί μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίες είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε εναλλακτικές λύσεις. Μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας μετά την τελευταία μεταρρύθμιση που έχει γίνει έγινε σαφές ότι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν χρηματοδότηση. Εδώ δεν ήμασταν απόλυτα σύμφωνοι. Εμείς θεωρήσαμε ότι όλα τα σχέδια για την αλία θα πρέπει να εξεταστούν βάσει της αξίας τους και όχι μόνο επειδή προωθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, μεγάλη τεχνολογική επένδυση τα σχέδια ιχθυοκαλλιέργειας και είναι πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν στα σχέδια αυτά χωρίς να έχουν καμία απόλυτα υποστήριξη. Αυτό είναι λάθος εκτίμηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Όταν μιλάτε για αυτόχθονα θαλάσσια είδη, δεν ξέρω αν θεωρείτε τον ερυθρόπτερο τόνο σαν ένα αυτόχθονο είδος. Στη Γαλλικία, παραδείγματος χάρη, έχουμε την ε, ανάπτυξη καλλιέργειας της ε, Ιαπωνικής πεταλίδας. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε, αν θα πρέπει να αναπτύξουμε και τέτοια είδη τα οποία δεν είναι απολύτω αυτόχρονα. Τέλος, για το θέμα των εισαγωγών, για το θέμα της εξέτασης των ε, τοξινών που μπορεί να υπάρχουν στα δίθυρα μαλάκια, η Κομισιόν έχει αλλάξει την χημική μέθοδο που χρησιμοποιείται προς το παρόν για τον έλεγχο και θεωρεί ότι είναι καλύτερη η νέα μέθοδος η οποία υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να εξετάσετε τη δυνατότητα τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την οδηγία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεχίσουν, παραδείγματο χάρη, οι τρίτε χώρε να χρησιμοποιούν παλιέ μεθόδου όταν εμεί έχουμε αλλάξει τη δική μα μέθοδο. Αυτό θα είναι αντιφατικό και θα οδηγήσει σε προβλήματα. Και πάλι σας λέω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση έναντι των εισαγωγών σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στην Κομισιόν και μετά στον κύριο Μιλάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, διότι η Κομισιόν επίσημα σε επίπεδο επιτρόπου θα αποφανθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί εκεί. Συμφωνώ τώρα και με τους ομιλητές. Συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή για τη διαπίστωση που κάνει, την οποία και συμμεριζόμαστε. Όμως όσον αφορά τις προτάσεις που κάνει στην έκθεσή του, ίσως υπάρξουν κάποιες αμφισβητήσεις από την πλευρά μας που θα εκφραστούν, θα διατυπωθούν αργότερα, όπως σας είπα, όταν η έκθεση θα έχει επίσημα ε, παρουσιαστεί στην Ολομέλεια. Οι σημερινές μου λοιπόν παρατηρήσεις δεν έχουν σαν αντικείμενο παρά μόνο να βοηθήσουν τον ε, εισηγητή να διευκρινίσει ίσως κάπως περισσότερο το περιεχόμενο της εκθεσής του. Πρώτα απ' όλα για το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την ανάπτυξη της θεατοκαλλιέργειας. Ξέρετε ότι δεν περιλαμβάνεται η πρόταση αυτή στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φετινό και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο. Το ίδιο όσον αφορά και για ένα ειδικό ταμείο για την υδατοκαλλιέργεια. Όπω και η κυρία Φράγκα, και εμεί πιστεύουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο σε μια εποχή που αναρωτιόμαστε κατά πόσο το σημερινό ταμείο θα διατηρηθεί στο μέλλον μετά τη μεταρρύθμιση των διευθυντικών ταμείων για το 2014 και μετά. Συνεπώ, αλλά και πάλι ε, αυτό που σας λέω είναι μια εκτίμηση που κάνω εγώ για να βοηθήσω τον εισηγητή. Τίποτα παραπάνω. Όσον αφορά την κατάρτιση τώρα, Ξέρετε ότι ήδη στις περισσότερες χώρες υπάρχει τέτοια κατάρτιση, ειδικά για όσους απασχολούνται επαγγελματικά στην υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχει τέτοια κατάρτιση λοιπόν επιπλέον από τη Γεωργία. Για το σημείο 4 τώρα του εισηγητή, εκεί αναφέρεται σε κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με το πιο σημαντικό διοικητικό εμπόδιο που έχουμε στην Ευρώπη για τις δατοκαλλιέργειες. Και αυτό είναι ο χώρος που χρειάζεται, ο εντοπισμό χώρων κατάλληλων για την ανάπτυξη της δατοκαλλιέργειας. Όπως και ο συγκεκριτής, έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι θεμελιώδες για να αναπτυχθεί η δατοκαλλιέργεια. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί περιορίζει το σημείο αυτό στις θαλάσσιες περιοχές ο συγκεκριτής, γιατί δηλαδή άλλες λεκάνες δεν ε, μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άρα ρητά να αναφερθούν στο εγγραφό του. Όσον αφορά τώρα τη διοικητική απλοποίηση, συμφωνούμε απόλυτα για να συνεισφέρουμε και εμείς στην μείωση της γραφειοκρατίας. Ξέρετε όμως ότι τα εμπόδια αυτά απορρέουν από τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για κείμενα τα οποία έχουν ε, υιοθετηθεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα η σήμανση για μια βιολογική υδατοκαλλιέργεια είναι μια ενδιαφέρουσα πιστεύουμε πρωτοβουλία και μάλιστα επειδή όπως ξέρετε η κοινότητα έχει αναπτύξει κανονισμό για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια που αποτελεί μέρος της βιολογικής γεωργίας. Οπότε εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι στο σημείο 7 ο εισηγητής αναφέρει την επέκταση του ορίου για, την, για αλλά τέτοια όρια υπάρχουν ήδη. Ο κοινοτικός κανονισμός για την υδατοκαλλιέργεια, τη βιολογική, υπάρχει, αλλά ίσως όχι στο βαθμό που θα το ήθελε ο εισηγητής. Τώρα για την έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχει ο τρέχον προπολογισμό, ο οποίος αφιερώνεται στην υδατοκαλλιέργεια και είναι σημαντικό στέκτο πρόγραμμα πλαίσιο περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ αφιερώνει στην έρευνα για την υδατοκαλλιέργεια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτό το βασικό εμπόδιο. Όπως και η κυρία Φράγκα, έτσι και εμείς δεν θέλουμε η έρευνα να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ντόπια είδη ή σε άλλα είδη είτε πρόκειται για την Γαλλία, είτε πρόκειται γενικότερα για την Ευρώπη. Και μιλάω για τη Γαλλία, γιατί στη Γαλλία έχουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα στρίδια, την καλλιέργεια στριδιών. Είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 8.000 ε, άνθρωποι επασχολούνται στον κλάδο. Και δεν είναι ντόπιο προϊόν, έτσι. Είναι μην, μη ντόπιο, αλλά που έχει προσαρμοστεί και έχει αφομοιωθεί στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Στο σημείο 9 τώρα. Λέτε, τα εισαγόμενα προϊόντα να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουμε στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν με τους τρέχοντες ε, κανόνες να πετήσουμε κάτι τέτοιο. Διότι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές απορρέουν από την εθνική πολιτική περισσότερο παρά από τη διεθνή. Για τους κορμοράνους ε, συμφωνούμε με την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τα ε, φτηνά αυτά να μην πλήττουν οικονομικά το κλάδο της ατοκαλλιέργειας. Αλλά για αυτή την προβληματική έχω μιλήσει και άλλη φορά. Δύο σημεία ακόμα. Πρώτον, θα θέλαμε ο εισηγητής του Κοινοβουλίου που δουλεύει για την υδατοκαλλιέργεια αλλά και για την ε, μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής φυσικά να συμπεριλάβει την υδατοκαλλιέργεια είναι μια προβληματική που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα και ελπίζουμε έτσι από το Κοινοβούλιο να έχουμε έναν προσανατολισμό ο οποίος θα είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη της μεταρρύθμισης αυτής της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Τέλος, υπενθυμίζω στον εισηγητή ότι είμαστε στη διάθεσή του για ό,τι πληροφορίες χρειάζεται. Όπως επίσης και για τα αποτελέσματα του Impact Assessment που έγινε όταν η Επιτροπή ετοίμασε τη στρατηγική της για την υδατοκαλλιέργεια. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μιλάνα περνάει ο χρόνο. Λοιπόν, για να είσαστε σύντομο λίγο παρακαλώ για να κλείσουμε τη συζήτηση. Τρία λεπτά μόνο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα επινετικά σχόλια. Μια δουλειά που εγώ θα έπρεπε να σα ευχαριστήσω και το κάνω και του βοηθού μου και τον ε, Δ. Κοαράντα τη Γραμματεία που συνεργάστηκα μαζί μου στενά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Συγχαρητήρια σε όλου με όσου συνεργαστήκαμε. Επίση σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, τα θετικά. Τρεις, τρία σύντομα σχόλια. Το θέμα της διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης όπου ψαρεύουμε το ψάρι στη θάλασσα, κάνουμε χθιάλευρα και το δίνουμε τροφή αυτό στι γελάδε. Και υπάρχει κίνδυνο να πάρουμε φυτικές πρωτεΐνες, α πούμε σόγια, και να δώσουμε στα ψάρια. Σω χρειάζεται μια καλύτερη ρύθμιση, καλύτερα τα ηχθάλευρα να τα δίνουμε στα ψάρια και να εκτρέφουμε τα θηλαστικά με προϊόντα της γεωργίας. Δηλαδή, να απλουστεύσουμε τους κανόνες. Το να θέλουμε σήμερα στην διατροφή να βάλουμε πρωτεΐνες που δεν προέρχονται από τα ψάρια θα πρέπει αναλογικά να μην δημιουργήσει πρόβλημα αλλά αντίστοιχα να επιτρέψει στα να τρώνε αυτά που συνήθως τρώνε. Αυτά για την διατροφή όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Δεύτερο, Συμφωνώ με την πρόεδρό μας. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι το μικρό είναι ωραίο. Αλλά το μικρό και ωραίο πολλές φορές δεν είναι κατά ανάγκη χρήσιμο στην οικονομία. Όταν έχουμε ψηλή συνιστόσα τεχνολογίας, θα πρέπει να πούμε ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται ενίσχυση. Εγώ λέω να οριστούν τα χαρακτηριστικά των μικρών και των μεγάλων, τα χαρακτηριστικά της παραγωγής να καθορίσουν την πρόσβαση στο ταμείο. Δηλαδή, αν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που την έχουμε ορίσει να υποστηριχθεί. Δηλαδή η επιλογή να μην γίνεται υποκειμενικά με βάση τον ετούντα, αντικειμενικά να κρίνεται, αν ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα έχουμε ορίσει. Όσον αφορά τα μη ντόπια ψάρια. Τα ντόπια ψάρια Σε αυτά μπορούμε να επενδύσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα, αλλά μην έχουμε αμφιβολίες. Πρέπει να γίνουν επενδύσει και σε μία αυτόχρονα είδη. Όπως γίνεται και στην κτηνοτροφία. Η γενετική επιλογή μερικών ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή ιστορικά έγινε μέσω διασταυρώσεων, βελτίωσης των ειδών προκειμένου να παράγουμε περισσότερο κρέας, περισσότερο γάλα, όλα αυτά είναι θεμητά. Αυτό πρέπει να γίνεται με βάση βιώσιμων παραμέτρων. Χωρίς αυτό να αποκλείει και τα μη αυτόχθονα είδη. Αυτό που έθεσε η Κομισιόν τώρα. Για το γλυκά νερά και τον χωροταξικό σχεδιασμό συμφωνούμε. Δεν συμφωνώ όμως με τον κανονισμό 710 της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Μεγάλη σιγή εκ μέρους της Κομισιόν. Το Κομισιόν δεν του δόθηκε δυνατότητα να πει τίποτα. Εγκρίθηκε τον Αύγουστο ο κανονισμός δεν τον αξιολογήσαμε εμείς, ούτε εμείς, ούτε το Κοινοβούλιο. Ο κανονισμός αυτός έχει όρια. Έχει μια συναισθηματική διάσταση για το βιολογικό γενικά. Άνοιξε μετά ένα μικρό κεφάλαιο για την υδατοκαλλιέργεια για να βολέψει όποιον θέλει να κάνει βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Εγώ θέλω να συμβιώνουν αυτά τα δύο εργαλεία έχουμε και βιολογική και βιομηχανική υδατοκαλλιέργεια. Η βιομηχανική μπορεί να έχει καλύτερη τύχη στην αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητες που να επιτρέπουν να εφαρμοστεί η πολιτική προώθηση καλής ποιότητας τον μη φαύλο κύκλο, όπως τον είπε ένας συνάδελφος. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιλάνα. Ε, περνάει ο χρόνο. Γρήγορα πάμε στο επόμενο σημείο, το 5 για την πράσινη βίβλο, γιατί έχουμε τι 5. Μετά έχουμε και τι ε, ποσοστό για τη Μεσόγειο. Προσοχή, πρέπει να φροντίσω να τηρώ και το χρόνο. Λοιπόν, έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε Πατράου και μετά θα έχουμε και τον κατάλογο των ομιλητών βέβαια που θα παρεύουν για το θέμα σα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. η Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει την ευθύνη συναπόφασης μέσα στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ο κύριος Κουέφ από την Προεδρία, τον οποίο ήδη ε, για την πρωτοβουλία αυτή και η Κομισιόν έχουν συμβάλει Προ την κατεύθυνση αυτή. Από την πλευρά τη Επιτροπής Αλία, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Κρέσπο, η οποία έχει συμβάλει ιδιαίτερα στην εκπόνηση αυτή τη έκθεση με μεγάλη αφοσίωση και μεγάλη προσπάθεια μου έχει δώσει μεγάλη βοήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου επίση, ιδίω του σκιώδει εισηγητέ, που ήταν απαραίτητοι συνεργατέ ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο αυτό το θέμα της κοινή πολιτικής αλίας και να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες του τομέα αυτού σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι παρόντες και θέλω να τονίσω ότι είναι εδώ παρόντες μια ομάδα από Πορτογάλους δημοσιογράφους από τις Αζόρες και αυτό δείχνει και ποιες είναι οι προσδοκίες που υπάρχουν από τη μεταρρυθμισμένη αυτή πολιτική αλίας όπως ελέγχθη στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων είχε τονιστεί ότι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε τότε ήταν πριν από την κατάθεση της έκθεσής μου στις 5 Νοεμβρίου και η οποία ακολούθησε μια κάπως σύντομη χρονική περίοδο αν σκεφτούμε τη σημασία αυτής της εργασίας αλλά επίσης και μια έντονη περίοδο εργασίας, όπου με τη βοήθεια των συνεργατών μου προσπάθησα να συμπιλήσω τις μελέτες διαφόρων οργανισμών για τα θέματα αυτά και να καταλήξω σε μια σύνοψη για τις εκθέσεις αυτές και να παρουσιάσω τις προσδοκίες τους για τα πιο σημαντικά θέματα που άπτονται της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και εδώ αναφέρομαι περισσότερο στο έργο των Συμβουλευτικών Περιφερειακών Συμβουλίων. Υπάρχει μια μεγάλη πολυπικιλία φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλίας και μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες του Τζο Μπόρτς που ήταν ο προηγούμενος Επίτροπος Αλίας. Οργανώσαμε δύο εργαστήρια που αφορούσαν αποκλειστικά λοιπόν τα θέματα αυτά της κοινή αλλιευτικής πολιτικής όπου ήταν παρόντες εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν, του Συμβουλίου, αλληλείς, ε, εφοπλιστές στον αλληλευτικό κόσμο, πολιτικοί, επιστήμονες κτλ. Η έκθεση λοιπόν αυτή η οποία έχει παρουσιαστεί από το ταπεινό μου άτομο δεν είναι απλώς προϊόν μονοφωνίας και προσωπικής άποψης, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας επαφής και της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό. Προσπάθησα λοιπόν έτσι να αφουγκραστώ τις ε, προσδοκίες και τα αιτήματα όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται στον τομέα αυτό σε σχέση με τη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Η έκθεση αυτή, επομένως, έπρεπε να ε, περιοριστεί και σε ένα συγκεκριμένο μήκος, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα αυτό θα έπρεπε να συνδυαστεί με την πλήρη κάλυψη όλων των θεμάτων, όλη τη θεματολογία που είναι παρούσα στο θέμα αυτό. Και επομένω προσπάθησα να συμπυκνώσω όλε τι γραμμέ μελλοντική δράση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρώ ότι είναι απαραίτητε. Αλλά πολλέ φορέ παρουσιάζοντά του με πιο απλοποιημένο και γενικό τρόπο από ό,τι απαιτούσαν. Και έρχομαι τώρα στην ουσία της έκθεση πέραν της ενσωμάτωσης της αξιολόγησης από, από μένα της πράσινης βίβλου, πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και ορισμένα έγγραφα τα οποία έχουν νομικό χαρακτήρα και επίσης είναι απαραίτητο να τονίσω ότι σε αιτιολογικές σκέψεις προσπάθησα να αναφέρω ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία διαμόρφωσαν την προβληματική αυτή για εμένα. Προσπάθησα λοιπόν να χωρίσω το εκτελεστικό κομμάτι αυτού του αυτή τη έκθεση σε δύο κομμάτα. Κομμάτια γενικά θέματα και ειδικά θέματα. Κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και την κατανόηση όλων. Το γενικό τμήμα αναφέρει κυρίως στις κύριες πτυχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη και που για μένα είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση. Ενώ το δεύτερο τμήμα που έχει να κάνει με τα επιμέρους στοιχεία καθορίζει ποιες θα πρέπει να είναι οι κύριες κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης, όπως τις προβλέπω εγώ και όπως τις ατενίζω αυτή τη στιγμή και όπως θεωρώ ότι θα πρέπει να προταθούν από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την άποψη αυτή <clears throat> καταγράφω πέντε βασικούς άξονες. Καταρχήν, η προστασία και η διατήρηση των πόρων και ε, επιστημονικές γνώσεις. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται εδώ να επανέλθω σε όλη την έκθεση που έχετε ενώπιόν σας και να σας την διαβάσω. Απλώς θέλω να τονίσω ορισμένες πτυχές της που μου φαίνεται ότι είναι οι πιο σημαντικές και είναι πιο ενδιαφέρουσες για την συζήτησή μας. Προστασία λοιπόν των πόρων και επιστημονική έρευνα. Εδώ θέλω να τονίσω τη σημασία να υπάρξει μια μεγαλύτερη επένδυση στην επιστημονική γνώση και έρευνα, γιατί η μεταρρύθμιση θα πρέπει να ακούει στα επιστημονικά πορίσματα της έρευνας για τους θαλάσσιους οργανισμούς και την αλία. Είναι θεμελιώδης λοιπόν η έρευνα και από εδώ και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε με μια μεγαλύτερη επιλεκτικότητα των τρόπων αλίας ώστε να αποφύγουμε τις υπερβολικές, τα υπερβολικά αλλιεύματα, αλλά να εξασφαλίσουμε αντίθετα μια αλία η οποία είναι όλο και πιο υπεύθυνη και εξασφαλίζει και την βιωσιμότητα των αλληλευτικών πόρων. Και ήθελα να τονίσω λοιπόν εδώ την ανάγκη να υπάρξει μια αυστηρή και εξαντλητική καταγραφή των χαρακτηριστικών μέγεθο, μεθοδιαλία κτλ. του τωρινού αλευτικού στόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χωρί κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προ αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και το οποίο θα καλύψει τι προσδοκίε όλων των εργαζόμενων στον τομέα αυτό. Δηλαδή είναι κεφαλαιόδηση, για να το κάνουμε αυτό μια διαφοροποίηση μεταξύ βιομηχανικού αλευτικού στόλου και βιοτεχνικού αλληλευτικού στόλου και φυσικά πρέπει να είναι σαφή τα κριτήρια τα οποία ισχύουν για τους δύο αυτούς τα δύο αυτά είδη αλληλευτικού στόλου και φυσικά τις διαφορετικές προδιαγραφές οι οποίες θα πρέπει να υπακούν. Δεύτερο σημείο είναι η αναγνώριση των προσόντων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αλλιών. Για μας είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αρχή ότι η αλία θα πρέπει να ασκείται με γνώμονα την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, απόδοση από τα αλλιεύματα. Μέσα σε αυτό θέλω να τονίσω πτυχές οι οποίες για μένα έχουν χαρακτήρα προτεραιότητες, δηλαδή να έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση των αλλιέων, την ε, αξιοποίηση της κατάρτισής τους, η κατεύθυνση των αλλιέων προς μια μεγαλύτερη χρήση του επιχειρήν στις δραστηριότητε τους, το να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όλοι οι αλληλείς βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, σε όλα τα κράτη και τα μέλη θα πρέπει να έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση, επίσης τις ανάγκες να εξασφαλιστεί η κοινωνική τους ασφάλιση, οι μηχανισμοί αρρωγής και χρηματοδότησης για τους ε, επαγγελματίες αλληλείς οι οποίοι μπορεί πολλές φορές να μείνουν με μειωμένα έσοδα ή και άνεργοι μέσω της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και επίσης, μέσα στο πλαίσιο αυτό του δεύτερου άξονα, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει μια πιστοποίηση, μια οικολογική πιστοποίηση ε, και μια σωστή κατεύθυνση των, ε, μια σειρά από οδηγίες προς τους ε, Τώρα έχουμε τον τρίτο άξονα που είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση και αυτό είναι ένα στίχημα. Να περάσουμε λοιπόν από μια κάθετη αντιμετώπιση σε μια οριζόντια αντιμετώπιση, κάτι το οποίο θα επιτρέπει μια πιο αποτελεσματική παρουσία όλων των επαγγελματιών του τομέα αυτού, με μεγαλύτερη δυνατότητα λήψης απόφασης από την πλευρά τους και τη δυνατότητά τους επίσης να επομιστούν μεγαλύτερες ευθύνες στους τομείς αυτούς σε ό,τι αφορά το καθεστώς διαχείρισης και θα μιλήσουμε μετά για τις ποσοστώσεις, είναι σαφές ότι για τόσο διαφοροποιημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τόσο διαφορετικούς τρόπους αλίες δεν μπορούμε να έχουμε μία πανάκια, ένα μοναδικό υπόδειγμα όπως αυτό των ποσοστώσεων και των ΤΑΚ. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις αναλλακτικές λύσεις, να μελετήσουμε τα τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτέ οι εναλλακτικέ λύσεις για να βρούμε ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση για κάθε συγκεκριμένη περιοχή και είδος αλίας. Τέταρτος άξονας, η υδατοκαλλιέργεια και τα μεταποιωμένα προϊόντα, τονίστηκε από τον κύριο Κουέφ, ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα χώρο για την υδατοκαλλιέργεια μέσα στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και επομένως η πτυχή αυτή προσπαθεί ακριβώς να εξασφαλίσει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο υπογραμμίζοντας πάντα τη σημασία που έχει η δατοκαλλιέργεια για την ανάπτυξη των παρακτήων περιοχών στις χώρες μας. Τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει όλο και περισσότερη έρευνα, ιδίω για την υπεράκτεια υδατοκαλλιέργεια και με στόχο να ενισχύσουμε όλο και περισσότερο την επιστημονική έρευνα ώστε η υδατοκαλλιέργεια να μπορέσει να μην είναι σε σύγκρουση με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Μία άλλη πτυχή η οποία έχει να κάνει με τις εξωτερικές σχέσεις και την ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτός ο πέμπτος άξονας, εξωτερικές σχέσεις. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παράγονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα αλίας, να επεκτείνεται δηλαδή η δραστηριότητα της αλίας σε άλλες περιοχές μέσω νέων συμφωνιών αλίας, αυτό για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα η ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το να κατανοήσουμε ότι ο τομέα αλληλεία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα από τομεακή έποψη και με τρόπο κατακαιρματισμένο, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια ευρύτερη πολιτική που είναι η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, λαμβάνοντα υπόψη και τι δυναμικότητε και το δυναμικό που έχει μια τέτοια πολιτική. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ευρύ πλαίσιο πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να εμβαθύνουμε περισσότερο ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα για τη μελλοντική πολιτική αλίας και αυτός είναι και ο στόχος μου. Όπως σας τόνισα προηγουμένως, προσπάθησα να λάβω υπόψη όλα αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία σε αυτή την έκθεση, αλλά πιστεύω ότι σε ένα έγγραφο αυτού του είδους είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν και να αντιμετωπιστούν σε πιο λεπτομεριακό επίπεδο όλα αυτά τα θέματα. Παραγωγή χάρη περισσότερε σε ό,τι αφορά τα θέματα εμπορία. Ακόμα και μία συστηματική αντιμετώπιση σε ένα ειδικό τομέα της έκθεσης, να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει εποπτεία και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αλληλείας με μια διαδικασία πιστοποίησης τόσο για την ιδιωτοκαλλιέργεια όσο και για την ελεύθερη αλληλεία, να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει μια αηφόρος μεταποιητική βιομηχανία για τα αλλιεύματα, επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα όπως οι συγκλίνουσες προσπάθειες για να μην υπάρξουν στρεβλώσεις, μια καλύτερη μορφή εποπτείας και ελέγχου, να υπάρξει επιπλέον η δυνατότητα να δώσουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στις υπερπεριφερειακές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου χρειάζεται πιο πολυθετική διάκριση, αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στον αλλιευτικό τομέα και πάλι με συγκεκριμένες μνήες των προβλημάτων που αντιμετωπίσουν ορισμένες περιοχές στη Βαλτική, στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ειδικά προβλήματα τα οποία και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αξίζουν περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη εμβάθυνση. Είμαι έτοιμη να δεχτώ τη συμβολή και των συναδέλφων και ελπίζω στη συνεργασία όλων των βουλευτών αυτής της Επιτροπής και ιδίως των σκιωδών εισηγητών με τους οποίους είχα την ευκαιρία με κάποιους από αυτούς να συναντηθώ την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και έχουμε ε, καθορίσει και νέε συναντήσεις στο μέλλον. Μας πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνος γιατί όλες οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 11ης Δεκεμβρίου. Γι' αυτό το λόγο ήδη εργαζόμαστε με μεγάλη ένταση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό δυνατό και φυσικά όταν έρθει σε ψηφοφορία αυτή η έκθεση τον Ιανουάριο θα πρέπει να γίνει αυτό ώστε να μπορούμε να είμαστε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Λοιπόν, ο κατάλογο των ομιλητών. Θα σα πω ποιοι είναι για να μην έχω ξεχάσει κανένα. Δύο λεπτό καθένα θα έχετε, έτσι. Δύο λεπτά. Dogs, Davis, Haglund, Lobin, Hackton. Για την ώρα, apuntada, ya está apuntada Ναι, ναι, σας έχω. Τότε την από την ώρα είπαμε και πότε τσεκ. Δύο λεπτά, αλλά μετράω, ε, Καπούλο Σάντος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας την κυρία Πατραουνέβη για την έκθεσή της και φυσικά έχω μια θετική αντιμετώπιση γιατί νομίζω ότι δίνει σωστές και αντικειμενικές απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η Κομισιόν στα πλαίσια της Πρασίνης ε, Βίβλου. Υπάρχουν σημεία βέβαια που έχω επιφυλάξει ή ακόμα και διαφωνίες και θέλω αυτά να τα θέσω υπόψη της κυρίας εισηγήτριας. Το πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά το υπόδειγμα των ποσοστώσεων. Εγώ εντυπωσιάζομαι ότι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη νη και στα σημεία 10 και 32, η, η υποστηρίζει αυτό το μοντέλο όπου δημιουργεί τόσες αντιδράσεις σε πολλές χώρες μέλη, όπως ακόμα και η δική μας χώρα, η Πορτογαλία. Υπάρχει αυτή η ανάγκη περιοδικών τροποποιήσεων για αυτό το σύστημα, αλλά το σύστημα της σχετικής σταθερότητος έχει εξασφαλίσει κάποια ισορροπία σε ένα τόσο δύσκολο θέμα. Δεν θεωρεί η συγγήτρια ότι η εγκατάλειψη του συστήματος των ποσοστώσεων θα ενισχύσει τις εταιρείε με μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό επίπεδο, θα ε, θίξει την αηφορία με την αύξηση των αλλιευμάτων. Δεν θεωρεί η συγγήτρια ότι ένα νέο μοντέλο, αν δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, αλίες, τις μορφές αλίες πολλαπλού χαρακτήρα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και αυτό αφορά ιδίως χώρες όπως είναι η Πορτογαλία. Και θέλω να θέσω τα εξή ερωτήματα στην εισηγήτρια. Βλέπω στα σημεία 4 και 11 της έκθεσή σας μία φαινομενική αντίφαση. Στο σημείο 4 μιλάτε σε υπερεπενδύσεις, εάν αυτό μπορεί να γίνει στην αλία, ενώ στο σημείο 11 λέτε ότι υπάρχει μία έλλειψη απενδύσεων σε ορισμένου τομεί. Μόνο μια τελευταία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Καλά, κλείνω αμέσω. Και για τα σημεία 31 και 34, νομίζω ότι η συγγήτρια με την πρότασή της κινδυνεύει να αφαιρέσει εξουσίες από το Κοινοβούλιο τώρα που έχουμε τις εξουσίες Τη συναπόφαση μου φαίνεται κάπω συγκεχημένη. Η διατύπωσή τη, αν μπορεί να τη διευκρινίσει καλύτερα, θα είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ για την επίκυριά σα. Η κυρία Ντότ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Τώρα, έχοντας μιλήσει στη Βόρεια Ιρλανδία με διάφορους αλείς, νομίζω ότι συμφωνούν με τις αρχές της διατήρησης των αποθεμάτων, τις αρχές που λέει να έχουν αξιοπρεπή ζωή οι αλείς και να είναι αποδοτική η αλία. Όμως, θα ήθελα να τονίσω και πόσο μεγάλη σημασία έχει η περιφερειοποίηση, η, αποκέντρωση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η προσέγγιση που έχει η σημερινή και ελευθερική πολιτική πρέπει να αλλάξει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ζητάω λοιπόν από την εισηγήτρια και την Επιτροπή μας να προσπαθήσει να δουλέψει πάνω σε, ένα, μια συνένεση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, σε συνεργασία με τον κλάδο, με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να πετύχει η πρόταση αυτή. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα όσον αφορά τη δικιά μου περιφέρεια. Η, η μιλάει για την πράσινη βίβλο και την υπεραλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα ευρύ θέμα. Στην Βόρεια Ιρλανδία έχουμε μειώσει από 220 τράτες σε 130 αλλιευτικά σκάφη τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχει δηλαδή τεράστια μείωση του στόλου μας και άρα και της αλλιεύσης. Οπότε εγώ δεν βλέπω να υπάρχει υπεραλίευση από εμά στην Ιρλανδική θάλασσα. Ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι εκείνο της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης που στηρίζει και θα στηρίξει ό,τι κάνουμε στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα έπρεπε να κοιτάξουμε και άλλα θέματα, όχι μόνο τα αποθέματα ή τις επιπτώσεις ε, στην θάλασσα. Επίσης, να προσθέσω και κάτι ακόμα. Αν θέλουμε εναλλακτική, αν κάτι άλλο δηλαδή εκτός από τα τάκ και την διαχείριση που έχουμε μέχρι τώρα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την σταθερότητα στους αλληλευτικούς πόρους και στη διαχείρισή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ανδρέας Βαρέα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό και υπάρχουν και τόσες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τα όσα μα είπε. Η έκθεσή της είναι πραγματικά μια έκθεση που έκανε πολύ γρήγορα προσπαθώντας να συμπεριλάβει τα πάντα. Αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αν και θα έπρεπε. Το θέμα τώρα των κριτηρίων προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια για την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτική μας και το κριτήριο της βιωσιμότητας της αλίας όπως ε, επίσης το θέμα της διατροφής από την αλία του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι πράγματα που σαφώς και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πολύ ενδιαφέρον μας φάνηκε το κριτήριό σας για την ε, αλληλευτική δραστηριότητα, πολύ θετικό και πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αναφέρεται η δυνατότητα αλλαγής των ε, αρχών της σχετικής σταθερότητας τα υποσωστώσει και τα τάκ τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Όπω επίση να αλλάξει το θέμα τη οικονομική βιωσιμότητα, το κριτήριο αυτό και τη αποτελεσματικότητα και τη ανταγωνιστικότητα. Όπω είπαμε και νωρίτερα, πρέπει να εκτιμήσουμε και την υπεραλίευση. Πόσο, πού και ποια είναι τα είδη τα οποία κινδυνεύουν. Μία ερώτηση έχω μόνο παρακαλώ, μια που δεν έχουμε χρόνο. Μια ερώτηση λοιπόν έλεγα για το σημείο 33 ο κοινοτικός οργανισμός ελέγχου της αλίας. Ίσως δεν μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα, αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβω. Πρόκειται για έναν σούπερ οργανισμό. Και μετά στο 32 που λέει για τη δημιουργία περιφερειακών αντίστοιχων οργανισμών. Πώς θα γίνει αυτό. Περιφερειοποίηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερο αυτή την ιδέα σας. Και κατά τα άλλα μου απαντήσατε για τις γυναίκες, εντάξει. Φαντάζομαι θα μου απαντήσετε κάποια άλλη στιγμή παρετέρω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια μας έδωσε μια χρήσιμη βάση δουλειάς. Τρία σχόλια. Πρώτον, έχουμε τεράστιες ποσότητες ψαριών που αλλιεύονται έξω από τα ύδατα της Ένωσης. Έχουμε μόνο το 8% του πληθυσμού μας αλλά η επίπτωση εκεί στη δράση ξεπερνάει πολύ τα, των ακτών μας. Για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αν ήταν εύκολο, θα το έχουμε φτάσει αυτό το επίπεδο. Χρειάζεται κόπος για να έχουμε μακροπρόθεσμο κέρδος. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ που βάζει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ως όριο θα πρέπει να αναγνωρίσει μια δύσκολη μεταβατική περίοδο. Τρίτο, η οικοσήμανση, οικολογική σήμανση. Φυσικά αυτό είναι σημαντικό. Παράλληλα με την κάλπ της Ένωσης προκειμένου να πετύχουμε βιωσιμότητα κάτω από τις σωστές συνθήκες, τα χρήματα θα πάνε στις τσέπες των ψαράδων. Με ένα πριμ στα ψάρια που αλλιεύουν, αλλά μη δημιουργούμε διπλές δομές. Πριν από 13 χρόνια, η Unilever και η WWF δημιούργησαν ένα όργανο σε σχέση με την αλληλεία που είναι το 70% της συνολικής παγκόσμια αλληλείας, θα φτάσει ήδη με το 10% για πιστοποιητικά, δίνει πιστοποιητικά. Είναι υψηλό επίπεδο ο οργανισμός. Για το οικολογικό σήμα Ας φροντίσουμε να μην είμαστε υπερβολικοί, να μην κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα, παράγγελα, με δύο δομές καταχώρησης. Ο κύριος Χάγκλουν. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων, συγχαίρω την εισηγήτρια. Πολύ καλή δουλειά. και γενικά συμφωνούμε με την έκθεση. Μερικές λεπτομέρειες τώρα. Προκειμένου να μπούμε σε πιο ειδικά σημεία. Καταρχήν αλληλεία μικρού μεγέθους, μικρής κλίμακας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερες προδιαγραφές λεπτομέρειες μάλλον, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η μικρού επίπεδου αλληλεία. Θα συμφωνήσω φαντάσουμε με τροπολογίες. Το πρόβλημα της υπεραλίευσης, υπερβάλλοντας στόλου. Θα πρέπει να είμαστε και εδώ πιο λεπτομερείς, να υπάρχει μια επιστημονική βάση για την αυτοδιαχείριση, πιο περιφερειακή δηλαδή μέθοδο εφαρμογής όσον αφορά την αλία. Καλά θα είναι να είμαστε λίγο περισσότερο σαφείς στο τελικό κείμενο. Τέλος, αρπακτική ηχθής, η ηχθιοφάγα, πτηνά, κορμοράνι κλπ. Θα θέλαμε να υπάρχει μια σαφής παράγραφος κείμενο και γι' αυτό. Για τα προβλήματα με τις φώκες, τους κορμοράνους και άλλα αρπακτικά είδη ηχθείων. Πάντως πιστεύω ότι θα βρούμε μια καλή λύση στο τέλος. Η κυρία Λοβέν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Συγγήτρια. Άριστη γνωμοδότηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το που διαφωνούμε. Συμφωνούμε σχεδόν με όλα. Έχανα ένα καλό κεφάλαιο για το μοντέλο διαχείρισης, την αποκέντρωση, την περιφερειακή διάσταση. Ό,τι μας προτείνεται είναι πολύ ωραία. Δύο λεπτομέρειες μόνο με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Τα σημεία 43 και 44. Εξωτερικές σχέσεις. Αυτό που λέτε στο κείμενο δεν είναι σωστό. Δηλαδή να ενθαρρυνθούν νέες συμφωνίες που θα επιτρέψουν περαιτέρω απασχόληση και μείωση της φτώχειας. Δεν συμφωνώ, διότι η Κομισιόν έχει αξιολογήσει πολλές από αυτές τις συμφωνίες και από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν αποδεικνύει αυτό που λέτε εσείς. Στο σημείο αυτό λοιπόν οι θέσεις μας διαφέρουν. Μετά, σελίδα 14. Λέτε για τα τρία πιο σημαντικά σημεία. Να φροντίσουμε να υπάρχουν επαρκή πόροι για την, τον εφοδιασμό. Έχετε τρεις στόχους, αλλά πρέπει να βάλετε προτεραιότητες, διότι η πράσινη βίβλος της Κομισιόν μας λέει ότι αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των στόχων, θα πρέπει να επιμείνουμε να τηρείται να αφορά η βιοπικιλότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τους αλληλείς. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έκθεση της κυρίας Πατράου Νέβες είναι σαν την πράσινη βίβλο. Μου αρέσουν μερικές πτυχές της έκθεσής του, άλλες λιγότερο. Εάν, όπως θέλουμε, πρόκειται να φτιάξουμε ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο λειτουργεί, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από την κοινή αλληλευτική πολιτική και να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα την προσαρμόσουμε για να προχωρήσουμε. Ο Επίτροπος ε, Μπότς μίλησε για μια εκβάθρον μεταρρυθμίση και εγώ συμφωνώ για μια τέτοια αντιμετώπιση. Αναφέρθηκαν σε ορισμένε περιπτώσει η υπερβολική, ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου. Κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το σύστημα τη υπερβολική αλληλευτική ικανότητα, αλλά ανησυχώ πολύ την ε, αντιμετώπιση της Κομισιόν για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η υπερβολική αλληλευτική ικανότητα μέσω μιας πιο, ε, κεντρο, μια, πιο επικεντρωμένες σε επίγειες δραστηριότητες ε, αλληλεία. Εγώ δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι η αποκέντρωση είναι απαραίτητη και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μνήμα της αποκέντρωσης και από την εισηγήτρια στην έκθεσή της. Αν θέλουμε λοιπόν να επιβάλλουμε σε όλους ένα κεντρικό μοντέλο και να δώσουμε απλώ ένα μικρό κατσαβιδάκι για να αλλάξει κανείς τους μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι επαρκές για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με μία αντιμετώπιση αποκέντρωσης και να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σύγκληση μεταξύ των παραμέτρων που ισχύουν σε διάφορες περιοχές για τις αποφάσεις διαχείρισης που θα πρέπει να πρετανεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να έχουμε πραγματικά ένα αποκεντρωμένο τρόπο διαχείρισης για τις ε, δραστηριότητες μικρής κλίμακος. Η άποψη που έχει η Κομισιόν μπορεί λοιπόν να μην λειτουργήσει πάντα σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα με μία πανάκια να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Ας αφήσουμε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τις συγκεκριμένες αλληλευτικές περιοχές να αποφασίσουν ποιε θα είναι οι μέθοδοι και όχι να τους επιβάλλουμε κάτι. Επόμενος ομιλητής. Συγχαρητήρια για την ακρίβεια στο κείμενό σας. Και με τη χρονική πίεση κάτω την οποία λειτουργήσατε. Πολύ σύντομα τώρα. Μιλάμε για αποκέντρωση, περιφερειοποίηση. Ο συνάδελφος μίλησε πριν από μένα και αυτός αναφέρθηκε σε αυτό. Πιθανότητα όμως ακόμα να μην έχουμε δώσει τον σαφή ορισμό. Τι σημαίνει η αποκέντρωση, η περιφερειοποίηση. Επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε το θέμα της περιφερειοποίησης και ταυτόχρονα κοινούς κανόνες για κάθε χώρα μέλος σε ένα ενιαίο πλαίσιο, θεωρώ ότι η συγγήτρια και όλοι μας θα πρέπει να φροντίσουμε τελικά αυτή η περιφερειοποίηση να μην μείνει μόνο στα λόγια, αλλά να υλοποιηθεί και στην πράξη. Και ένα ακόμη, και κάνω έκκληση και προς την Κομισιόν, για τροπολογίες μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, ότι η πράσινη βίβλος θα είναι το μεγάλο θέμα για την Επιτροπή μας. Γιατί η πολιτική αλίας ειδικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία αρχίζει να ισχύει από αύριο το πρωί, μας βάζει μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία σε σχέση με το 2002. Δεν έχουμε χρόνο. Κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όμως την Κομισιόν, να μας δώσει λίγο χρόνο παραπάνω για να το δούμε καλύτερα το θέμα, το πρόβλημα μερικές βδομάδες ακόμη, όχι μήνες, βδομάδες. Να το μελετήσουμε καλύτερα και η δουλειά να είναι ακόμα πιο υποφελής. Ο κύριος Γκόρμπατσεκ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά να πετύχει συνένεση μεταξύ όλων των τομέων και περιφερειών της Ένωσης, προκειμένου να συνταχθεί η πράσινη βίβλος. Κάτι που αναφέρθηκε ήδη, αλλά το λέω κάτω από διαφορετικό φωτισμό. Επιστημονική έρευνα. Που συνήθως την αναφέρουν οι συγητές, αλλά πολύ συχνά αναφέρουν και την έλλειψη αντικειμενικών δεδομένων, επιστημονικών δεδομένων εννοώ. Αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση για μελλοντικό προγραμματισμό, προκειμένου Φερρυπίν να μειωθεί ο, ο υπερβάλλον στόλος. Γιατί αν πάρουμε στοιχεία που δεν είναι αξιόπιστα ή είναι απλώς εκτιμήσεις, σχετικά με τα αποθέματα Φερρυπίν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του στόλου χωρίς λόγο. Όπως έγινε με τη Ρέγκα στη Βαλτική. Πρόσφατα ακούγαμε ότι όλα είναι πολύ ωραία με τη Ρέγκα και έπρεπε να μειωθεί ο στόλος κατά 40%. Με βάση αυτό που είπε πριν από μένα ο κύριος Αντινόρο, αυτή η περιφερειοποίηση θα πρέπει να στοχεύει στην προστασία το βραχίας απόστασης αλίας μας. Αν το 80% είναι βιομηχανική αλία, τότε αυτή η βραχίας απόστασης αλία θα πρέπει και αυτή να προστατεύεται. Ο κύριος Μιλάνα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. θετική η θέση της συναδέλφου εισηγήτριας, ισορροπημένη. Το κεφάλαιο που συνδέεται με την υδατοκαλλιέργεια και την δουλειά που κάνουμε συνδέονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Πλήρης ακολουθία σε αυτά τα δύο. Μακάρι όμως να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί αυτή η έκθεση είναι σημαντική θα πρέπει να αξιολογήσουμε και εμείς, αλλά θα πρέπει να έχουμε περιθώριο να τη συζητήσουμε μεταξύ μας. Έχουμε ένα νέο επίτροπο για τα θέματα αυτά. Ίσως υπάρχει δυνατότητα να μας δοθεί και μας περισσότερο χρόνος. Ενδεχομένω να μην πάει στην Ολομέλεια αντί του Ιανουαρίου, να πάει το Φεβράριο. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό χρειάζομαι μονάχα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και από τη δική μου πολιτική ομάδα και νομίζω ότι θα είναι σημαντική η συμβολή μας. Και έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο και πάλι τονίζω και πάλι την ανάγκη της χωροταξικής αντιμετώπισης για την παράκτη, αλληλεία και η υδατοκαλλιέργεια. Είναι απαραίτητο να τονιστεί αυτό το στοιχείο για μένα και νομίζω ότι εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσουμε ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, η Κομισιόν μπορεί αύριο να επανέλθει εφόσον θα έχουμε την ακρόαση και να εκφράσει την άποψή τη για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πατράου Θέλω να πω μονάχα το εξή όμω προηγουμένω. Αν θέλουμε το θέμα αυτό να είναι έτοιμο για το Φεβρουάριο στην Ορομέλεια και αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε αρκετό χρόνο ώστε η Κομισιόν να λάβει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι απαραίτητο να κλείσει στι 11 Δεκεμβρίου η προθεσμή για τι τροπολογίε. Γιατί έτσι θα έχουμε μεταφρασμένε τι τροπολογίε μέχρι τι 14 Ιανουαρίου και θα έχουμε τι 12 μέρε που είναι απαραίτητε για συμφωνίε μεταξύ των πολιτικών ομάδων με μεταφρασμένε τροπολογίε, γιατί αλλιώ θα έχουμε πρόβλημα. Σα παρακαλώ λοιπόν <clears throat> όλου να λάβετε υπόψη ότι είναι σημαντικό το πρόβλημα της μεταρρύθμισης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν πρέπει να αλλάξουμε την ημερομηνία του Φεβρουαρίου για την Ολομέλεια. Και έτσι δεν θα χρησιμοποιηθεί πραγματικά η άποψη του Κοινοβουλίου. Δίνω το λόγο για πέντε λεπτά το πολύ στην κυρία Πατράου και μετά θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της Μέσης διάταξης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην καταδαπανίσω αυτά τα πέντε λεπτά. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Μπορώ να πω συνθετικά το εξή ότι υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο από παρατηρήσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί και ουσιαστικά είναι εκκλήσεις για να αναπτυχθούν περισσότερο στοιχεία τα οποία ήδη βρίσκονται δυνητικά στην έκθεσή μου. Εγώ συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομεριακή αντιμετώπιση και ανάπτυξη των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή και επίσης για να δώσουμε μια απάντηση σε ορισμένε παρατήρησεις οι οποίες έχουν διατύπωθεί που τονίσουν ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε μονάχα σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αντίθετα θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο και να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μεγαλύτερη ανάπτυξη και εξέταση σε λεπτομέρεια σε ορισμένα θέματα. Αυτό είπαν οι περισσότερε ερωτήσεις και θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να καλύψουμε τις ανησυχίε σα στο θέμα αυτό. Ένα άλλο σύνολο από παρατηρήσει είχε με διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσει το θέμα της αποκέντρωσης ή της περιφερο... περιφερειοποίησης. Ή πάρα πολλά από τα ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν ίσως διαφορετικά, τελικά καταλήγουν σε μια τέτοια προβληματική. Για τα θέματα αυτά εγώ πιστεύω ότι οι αμφιβολίες οι οποίες διατυπώθηκαν μπορούν να ξεπεραστούν με καλύτερη και επακριβέστερη διατύπωση στο έγγραφο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η βασική μου ιδέα ήταν να προσπαθήσω να εξασφαλίσω μια ισορροπία μεταξύ αυτού που είναι πραγματικά μια κοινή πολιτική αλίας με κοινέ προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών. <clears throat> Συγχρόνως όμως και μια ευέλικτη πολιτική αλεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι ιδιαιτερότητε και τι ειδικέ ανάγκε κάθε περιοχή και κάθε είδου αλεία. Περιλαμβάνουμε λοιπόν εδώ πέρα διαφορετικά υποδείγματα διαχείρισης των αλλιευτικών πόρων. Ενδεχομένως και μεικτά μοντέλα διαχείρισης περιλαμβάνονται σε μια τέτοια προβληματική, καθώς και η αρχή της ε, σχετικής Σχετική σταθερότητα, όπως αναφέρθηκε, κανείς δεν έχει διατυπώσει μια αντίθετη γνώμη στις ακροάσεις. Όλοι είπαμε ότι χρειάζεται αυτή η σχετική σταθερότητα, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στις τωρινές συνθήκες. Επίσης, σε σχέση με αυτήν την τριλογία που αναφέρω στη σελίδα 13 του εγγραφού, είναι πολύ σημαντική, τονίζουν ορισμένοι ότι, ρωτούν ορισμένοι μάλλον, ποια είναι η ιεραρχία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ αυτών των τριών σημείων. Εγώ νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να μην υπάρχει πραγματικά ιεραρχία, να συνδυάσουμε το κοινωνικό, το οικονομικό και το περιβαλλοντικό στοιχείο σε ίσο επίπεδο, ώστε όταν ένα από τα τρία στοιχεία βρίσκεται σε κίνδυνο να υπάρξουν διαφυλάξεις, μηχανισμοί διαφύλαξης, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών στοιχείων. Και τώρα, σε ένα τελευταίο λεπτό, θα ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ε, συνάδελφό μου, το συνάδελφο Καπόλας Σάντους, που έκανε την πρώτη παρέμβαση από την πλευρά των ομιλητών εδώ, λέγοντας ότι υπάρχουν ασυνέχειες, ελλείψεις συνοχής και έλλειψη γνώσης του τομέα αυτού. Βέβαια, έφυγε ο κύριος Καπόλας Σάντος, αφού έκανε την παρέμβασή του. Εγώ είμαι νεοφερμένη βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εγώ θέλω να υπάρχει πραγματικά διάλογος με του βουλευτέ. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια επίκριση, θέλω να έχω την ευκαιρία διαλόγου, την ευκαιρία να απαντήσω. Εγώ συζητώ πάντα με τους σκιώδει συγητές και θέλω να έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση. Διαφωνούμε να αναζητήσουμε τη λύση. Συμφωνούμε να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη λύση. Τώρα, όταν κάποιο είναι απόν στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δε, απόν στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων από στα εργαστήρια που κάνουμε στην Πορτογαλία, να έρχεται κάποιος να κάνει κριτική και μετά να μην είναι παρόν για να απαντήσει εγώ, ακόμα και σαν νέα βουλευτής σε αυτό το κοινοβούλιο, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτή είναι η καλύτερη συμπεριφορά. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας το τονίσω. Κοιτάξτε, μου είπε ότι είχε μια πήγουσα συνεδρίαση στη Γεωργία, έτσι νομίζω ότι μου είπε και γι' αυτό ήθελε να πάρει πρώτα το λόγο. Εδώ είναι όμως η βοηθός του η οποία σημειώνει τα όσα είπατε την απάντηση. Εγώ απλώς σας το λέω, ε, ως πρόεδρος προσπαθώ να είμαι ελαστική. Ο κύριος Καπούλα όντως μου το είπε ε, και γι' αυτό έφυγε, μου το είπε. Δεν είναι δικαιολογία, απλώς ό,τι μου είπαν ως πρόεδρο σας το μεταφέρω. Από εκεί και πέρα εσείς φυσικά είσαστε ελεύθεροι να μην συμμεριστείτε την δικαιολογία αυτή για την απουσία του κ. Καπούλα Σάντος. Στην περίπτωση αυτή τονίζω ότι είμαι πάντα στη διάθεση του κυρίου Καπόλα Σάντο για να συναντηθούμε διμερώ και να επιλύσουμε τα θέματα αυτά. Είναι Σίγουρα η βοηθό του που είναι εδώ παρούσα θα φροντίσει να του τα μεταφέρει όλα αυτά. Ωραία. Αύριο είπαμε έχουμε την ακρόαση. Η ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου. Σας είπα είναι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, φροντίστε να την τηρήσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω στις μεταφρασμένες τροπολογίε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε. Έχει κλείσει το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Δεν την ακούμε. Ο κύριος Ριμπελίνη δεν θα είναι εδώ σήμερα και μονέθεσε μένα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο και γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Λοιπόν, η έκθεση αυτή, όπως το έχουμε ήδη πει, είναι πρόταση της Επιτροπής που έχει να κάνει με μια μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο συστάσεων που γίνονται σε έναν περιφερειακό οργανισμό Αλίας που είναι η Γενική Επιτροπή Αλίας για τη Μεσόγειο. Ο κύριος Ριμπελίνη εξέτασε την πρόταση της Κομισιόν και συμφωνεί με τις συστάσεις που έγιναν από το Γενικό Συμβούλιο Αλίας για την Μεσόγειο και δεδομένου ότι το θέμα αυτό θα περάσει σε συναπόφαση επίσης, ο κύριος Ριμπελίνη έχει προτείνει διαγραφή του άρθρου 28 που αναφέρεται στην Επιτροπολογία. Αύριο, ξέρετε, αρχίζει να ισχύει η Λισαβόνα. Η Επιτροπολογία λοιπόν ως είχε μέχρι τώρα εξαφανίζεται. Και ανταυτής έχουμε τα άρθρα 290 και 291. Συνεπώς, ο κύριος Ριμπελίνη ε, διαγράφει το άρθρο για την επιτροπολογία και επαφίεται στα νέα άρθρα της συνθήκης. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ με τη δικιά μου έκθεση. Συνεπώ, κατά τα άλλα, η έκθεση αυτή δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο το θέμα τη επιτροπολογία ήταν και ελπίζω ότι κανένα από εσά δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα με την έκθεση αυτή. Από πλευρά τη Κομισιόν, αν δεν θέλει κανένα από εσά το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντονατέλα. Μήπω έχει κάτι να προσθέσει. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Άκουσα προσεκτικά την παρουσίασή σας όπως παρουσιάσατε δηλαδή το σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ομολογώ ότι εμείς δεν βλέπουμε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί μας επιτρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή πολύ γρήγορα αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στα πλαίσια της Γενικής Επιτροπής Ελίας για τη Μεσόγειο και που έτσι πολύ γρήγορα μπορούν να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο για να αποφύγουμε προβλήματα ερμηνείας και έτσι οι αποφάσεις αυτές να είναι περισσότερο ορατές. Πέρα από αυτό όμως η Επιτροπή θέλει να διατηρήσει και μένει στην πρότασή της. Θα έχουμε φαντάζομαι την ευκαιρία να ξανασυστήσουμε με την Επιτροπή σας και με τους συναδέλφους του Συμβουλίου. Αυτά έχω να πω προς το παρόν για αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ναι, σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για επιτροπολογία και για τα άρθρα 290 και 291, κυρίως γιατί πιστεύω ότι η Επιτροπή θα ετοιμάσει μία ανακοίνωση ακριβώς για τις πράξεις αυτές. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο σίγουρα που οι εισηγητές θα πρέπει να διαχειρίζονται την έκθεσή τους όσο γίνεται καλύτερα, χωρίς να έχουν όμως κάποιο μοντέλο για να ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Τι να γίνει. Και γι' αυτό ακριβώ είπα ότι το κύριο πρόβλημα ήταν το πρόβλημα της επιτροπολογίας εντό αγωγικών, και πώς θα το λύσουμε σε αυτό το διάστημα του ενός ή δύο μηνών μέχρι να έχουμε την ανακοίνωση. Ο κάθε εισηγητής με το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να δει πώς θα λύσει ό,τι προβλήματα επιτροπολογίας τίθεται με τα άρθρα 290 και 291 όπως σας είπα. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Παρακαλώ, ο κύριος Αρσένης. Arsenis, perdone, o για ya me confundo con todos los nombres griegos, de antes y después. Arsenis, perdone. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ε, είναι ένα πάγιο θέμα το οποίο μπαίνει πιο δυνατά με το, τώρα με τη συναπόφαση μετά τη Λισαβόνα το θέμα δηλαδή αν και το κομιτόλης θα περνάει μόνο από την Κομισιόν ή θα περνάει από το Κοινοβούλιο. Προφανώς και σε γενικές γραμμές ε, θα ρίνουμε πάντοτε να ε, εμπλέκεται όσο δυνατόν το περισσότερο το Κοινοβούλιο ε, στις διαδικασίες αυτές ε, για να αγγιάται ακριβώς και ότι ο λόγος των πολιτών της Ευρώπης θα ακουστεί. Ε, σε αυτή την ειδική περίπτωση ίσως η Επιτροπή να έχει δίκιο και ο λόγος είναι ότι ε, μιλάμε για ένα κείμενο το οποίο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει τη συμφωνία να το υιοθετούμε ω έχει. Είναι μια τυπική διαδικασία και είναι μια τυπική διαδικασία η οποία καθυστερούμε πάρα πολύ. Ε, σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε στο τέλος του 2009 για την απόφαση, ε, για την ε, που πρέπει να ενσωματώσουμε από το 2008. Και ούτε καν έχουμε ενσωματώσει, ούτε έχουμε καν ξεκινήσει τι αποφάσει του 2009 που πρέπει να ενσωματώσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ε, οπότε θεωρώ ότι ίσως ε, σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε απόφαση ε, λάβουμε η οποία μας επιταχύνει τις διαδικασίες να είναι η βέλτιστη. Ευχαριστώ πολύ. Permíteme, señora Senis, Κύριε Σένη, να σας εξηγήσω. Η ενσωμάτωση γιατί η πρόταση έγινε από την Επιτροπή όταν έγινε, πριν από ένα-ενάμιση μήνα. Δηλαδή, δεν φταίει το Κοινοβούλιο μας. Δεύτερον, οι συστάσεις του Γενικού Συμβουλίου αλία για την Μεσόγειο πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη, γιατί σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, τότε είναι συμβαλόμενα μέρη τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι διαφορετικό από την ΑΦΕ κλπ. Οπότε, ενώ εδώ δεν γίνεται καταπηγόντως η ενσωμάτωση, οι συστάσεις είναι υποχρεωτικές για όλες τις χώρες μέλη. Εντάξει, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κοινοτικό δίκαιο. Αν υπάρχει, ε, λέτε, νομικό κενό, δεν υπάρχει, γιατί είναι υποχρέωση για όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Επιμένω, το Γενικό Αυτοσυμβούλιο Αλίας για τη Μεσόγειο έχει μέλη που είναι συμβαλόμενα μέρη τη σύμβαση. Άρα έχουν την υποχρέωση. Έπειτα, δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί τίποτα άλλο, γιατί αρχίζει αύριο να ισχύει η Λισαβόνα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να συμμορφωθούμε με τις συνθήκες. Η επιτροπολογία είναι το μόνο πρόβλημα. Δεν είμαστε κατά τη ουσία τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με τι πτυχέ τη επιτροπολογία διαφωνούμε, που έχουν αλλάξει με τη Λισαβόνα και τώρα έχουμε τα άρθρα 290 και 290 ανταυτή. Ακόμα και αν θέλαμε, νομικά, ε, σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην νέα συνθήκη, εντάξει, καταλάβατε. Καταλάβατε αυτό σα λέω Έχετε κάποια αφιβολία. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σα μείνει αφιβολία. Προσπαθώ να σα το εξηγήσω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο Ριμπελίνη βέβαια, αλλά προσπαθώ να σα εξηγήσω το γιατί. Γιατί ο εισηγητή ε, προτείνει αυτό που προτείνει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσαρμοζόμαστε στη νέα συνθήκη που αρχίζει να ισχύει από αύριο και οι συστάσεις του Συμβουλίου πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή γιατί είναι συμβαλόμενα και τα κράτη-μέλη εκτός από την ευρωπαϊκή κοινότητα στην συνθήκη αυτή, στην, στο Συμβούλιο αυτό για τη Μεσόγειο. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή ανεξαρτήτως αν ε, τα κράτη-μέλη καθένα ξεχωριστά υιοθετεί και, και εφαρμόζει τις αποφάσεις όπως είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο έχει υποχρέωση να υιοθετεί εγκαίρως και να εφαρμόσει θεωρώ ε, σημαντικό να εγγυηθούμε ότι ε, αυτές οι διαδικασίες θα επιταχυθούν και θα φτάσουν, θα, θα αποκατασταθούν σε ένα επίπεδο αξιοπρέπεια, που σημαίνει ότι το 2009 θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει ή να έχουμε σωματώσει το 2009 και ούτω καθεξής και όχι να περνάνε ένα και δύο χρόνια. Και πραγματικά ε, εφόσον ε, έτσι και αλλιώ ε, οποιαδήποτε συζήτηση για το κομιτόλογι δεν έχει σημασία γιατί θα λυθεί από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γιατί έτσι και θα τα λύσει η συνθήκη της Λισαβόνας και τα λύνει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, είπα όμω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε για την προσαρμογή αυτή. Η Λισαβόνα λέει πώς πρέπει να έχουν τα πράγματα. Το πώς θα προσαρμοστούμε εμείς πρέπει να το κάνουμε και πρέπει κατά περίπτωση να φροντίσουμε για την προσαρμογή αυτή μέχρι να ετοιμάσει την ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να λέει ότι οι πράξεις αυτές και αυτές θα ακολουθήσουν το εξή μοντέλο. Ένα μοντέλο για να μπορέσουμε χωρί προβλήματα να συνεχίσουμε. Προ το παρόν δεν την έχουμε την ανακοίνωση αυτή τη Επιτροπή, γι' αυτό και πρέπει κατά περίπτωση να δούμε πώ θα προσαρμοζόμαστε στη Λισαβόνα. Άμα θέλετε, το συζητάμε. Εγώ το έχω μελετήσει πάντω και έχω προσπαθήσει να το καταλάβω. Πάντω, άμα θέλετε ευχαρίστω να συζητήσουμε κάποια στιγμή για να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που θέλω εδώ να προσθέσω είναι ότι εμείς δεν το κρίναμε πιο νωρίς αυτό, γιατί την πρόταση του κανονισμού δεν μας την είχε προτείνει η Επιτροπή. Και εμείς πολλά χρόνια πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέμε ότι η μεταφορά στο κοινοτικό δίκαιο των ε, συστάσεων της Επιτροπής για τη Μεσόγειο πρέπει να γίνονται γρήγορα. Όταν εκείνοι αργούν να ζητήσουν από εμά γνωμοδότηση, εμείς τι άλλο να κάνουμε. Είναι ένα παλιό ζήτημα αυτό, παλιό θέμα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι, κάθε άλλο. Εντάξει, δεν λέω ότι θα τα βάλουμε τώρα με την Επιτροπή, γιατί η Επιτροπή τι λέει, λέει ότι δεν έχει αρκετό προσωπικό, δεν έχει πολλέ δυνατότητε για να προχωράει πιο γρήγορα. Οπότε τι να κάνουμε, τέλο πάντων. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι τελικά η Αλία είναι πάντα η τελευταία ρόδα του κάρου. Τι να γίνει. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσιας διάταξης Έχουμε 10 λεπτά. Είναι η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προτινόμενων για το 2010 ε, συνόλων επιτροπωμένων αλλιευμάτων και ποσοστώσεων. Ο κύριο Πάτερσον από την Επιτροπή θα μα το παρουσιάσει. Παρακαλώ κύριε Πάτερσον. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομο. Και επειδή το θέμα είναι περίπλοκο, ζητώ συγγνώμη, γιατί θα είμαι κάπω επιφανειακό στην παρουσίασή μου. Οι βασικέ αρχέ. Η πρώτη είναι για εγκονισμό του Συμβουλίου για 140 τίτλοι. 145 τάκ, 3, 47 αλλιευτικές ευκαιρίες με διαπραγματεύσεις με τα παράκτια κράτη, 3 συστήματα περιορισμού των ε, προσπαθειών, Φέτος έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν έχουμε τεχνικά μέτρα, αλλά δεν έχουμε διεθνή μέτρα ΤΑΚ. Η αξία των αποθεμάτων, των αγγευμάτων, είναι 5 δις πέρυσι. Σας θυμίζω τους στόχους της ΚΑΛΠ. Βιώσιμη βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Κίνητρα για εξαγωγές. Η αρχή της σύνεσης, precaution, να ελαχιστοποιηθεί αρνητικές επιπτώσεις στα θεράσια συστήματα και μια καλή διαχείριση του συστήματος. Άλλοι στόχοι είναι να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα και των Αγγλίων και των καταναλωτών. Τώρα πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Κομισιόν για τη μεθοδολογία. Ευκαιρίες για το 2010. Πώς θα γίνεται η δειγματοληψία και ο έλεγχος. Έχουμε ε, στοιχεία από τις συμβουλευτικές επιτροπές και επιστημονική και τεχνική επιτροπή για την Αγγλία. Όπου υπάρχουν ε, μακροχρόνια προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν πρέπει να ορίζονται ευκαιρίε οι οποίε πάνε πέρα των δεσμεύσεων του Johannesburg ε, με βάση το 2015. Δεν πρέπει να κινούμαστε συστηματικά προ το στόχο αυτό. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου, αλλά δεν πρέπει και να κινούμαστε εναντίον τη απόφαση αυτή, τη συμφωνία αυτή. υπόψη ε, πολύ την αρχή τη όφρονα δράση και να έχουμε σταθερότητα. Περιορίζουμε αλλαγέ στα ΤΑΚ όσο περισσότερο γίνεται. Πώ γίνεται αυτό. Μία ταξινόμηση των αποθεμάτων ανάλογα με τι κατηγορίες και τις πληροφορίες και να εφαρμόζουμε σταθερού κανόνες. Χρειαζόμαστε σταθερούς κανόνες έτσι ώστε να πετυχαίνουμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα σε όλα τα μέρη τη Ένωση. Αυτό το διάγραμμα, το σχήμα το συζητάμε με τους αρμόδιους του, του, του κλάδου. Δεν θα γίνει πλήρη αναθεώρηση βέβαια τη ε, ΚΑΛΠ τώρα θα ήθελα να αναφέρω μερικά επιμέρους σημεία. Καταρχήν, τα αποθέματα που αξιολογήσαμε ως υπεραγγευόμενα ή με βάση την, τον βιώσιμο στόχο. Πολλά αλλιεύματα υπεραγγεύονται, αλλά η αναλογία των αλλιευμάτων έχουμε βελτίωση του βιώσιμου ποσού. Δεύτερο μέτρο. Πόσα αποθέματα μας λένε ε, οι ειδικοί ότι πρέπει να έρθουν στο μηδέν. Ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Προς τα τελευταία χρόνια είχα μία μικρή μείωση στις χειρότερες περιπτώσεις των αποθεμάτων. Ιδιαίτερα ένα ε, απόθεμα είναι ο βακαλάς της Βόρειας Θάλασσας. Η μπλε γραμμή δείχνει το μέγεθος των αποθεμάτων, η κόκκινη γραμμή δείχνει τους στόχους. Για την βιώσιμη αλληλεία, αυτή η κόκκινη γραμμή που είναι κάτω εκεί που σας δείχνω. Κινηθήκαμε προς τη γραμμή αυτή από το 2000 μέχρι σήμερα με ειδικά μέτρα για προστασία των αποθυμάτων του Βακαλά. Δυστυχώς την τελευταία χρονιά είχαμε αντιστροφή. Σε όρους βιομάζας είναι λιγότερο το ποσό σε σχέση με τον Βακαλάο. Μερικοί λένε ότι έγινε ανάκαμψη στο απόθεμα του κοντ αυτού του Βακαλάου. Του γάδου, του Εδώ μιλάμε για ψάρια που έχουν γεννηθεί το 2005. Μετά, την, μετά το έτος αυτό δεν έχουμε μεγάλο απόθεμα. Τα άλλα αποθέματα θα πρέπει να τα καλύψω πολύ γρήγορα. Θα μεγάλη αύξηση στο ΤΑΚ για την ΡΕΓΚΑ. Για τα άλλα αποθέματα στον πίνακα αυξήσεις. Νότιο Καλαρία. Καλαρία, γλώσσα. Στον κόλπο του Βυσκαϊκό και τον Βακαλά του Βορρά. Μειώσει στα τάκ. Μεγάλη μείωση στον spare dog. Μεγάλη μείωση για καλαρία δυτικά της Σκοτίας. Πιο μικρές μειώσεις για τη γλώσσα στην Ανατολική Μάχη. Νέρφοψ στην Ιρλανδία, Καραβίδα, Γάδο, Πατραχόψερο, Βακαλάο Μερλούκιο. Τελίκα. Η συμβουλή του είναι να μην γίνει αργία. Η Κομισιόν προτείνει μείωση μόνο 25%. Για 49 λεπτά έχουμε μείωση 15% με βάση τις υποστημονικές συμβουλές και 19 τάκ παραμένουν αμετάβλητα. Εδώ έχετε περισσότερες πληροφορίες για τα αποθέματα. Αυτά γρήγορα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Κοιτάξτε, χρόνο δεν έχουμε για να το συζητήσουμε ευρέως το θέμα. Έχω βρει πράγματα που δεν μου αρέσουν εδώ και ένα από αυτά είναι το θέμα του Μερλούκιου της Βόρειας Θάλασσας, όπου μιλάμε για 55.000 τόνους και έχει αλλάξει η πρόταση σε 46.300 κάτι, πολύ κάτω τέλος πάντων από αυτό που προτείνει η ΣΕΠ. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο ανάκαμψης και όταν μιλάτε για 20% μείωση, είναι για να πετύχουμε αυτό που εσείς έχετε προβλέψει στο σχέδιο διαχείρισης. Συνεπώς, τι να πω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και δεν καταλαβαίνω και την αιτιολόγηση. Γιατί σε ένα τομέα ο οποίος έχει πετύχει τους στόχους βιομάζας, εθνισιμότητας, το βρίσκω υπερβολικό το 20%. Έπειτα, ε, δεν νομίζω ότι μπορείτε να πείτε τα ίδια όταν έχουμε είδη τα οποία συνδέονται με ψάρια άλλα τα οποία έχουμε μιλήσει για διαφορετικά ποσοστά μείωσης. Υπάρχουν πολλά πράγματα εγώ που δεν έχω καταλάβει πάντως. Χρόνο δεν έχουμε γιατί πρέπει να συνεδριάσουν οι συντονιστές. Αλλά πολύ θα ήθελα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος βουλευτής να ρωτήσει κάτι τώρα, να μιλήσει, παρακαλώ. Και μετά θα κλείσουμε, έτσι, η κυρία Τόρτσου και ο κύριος Ρότσου. Και μετά κλείνουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που είχαμε, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπής μας και της Κομισιόν στο θέμα της περιοχής 7 και των καραβίδων. Οι καραβίδες είναι ένα από τα βασικά προϊόντα που αλλιεύονται από τους ε, αλληλευτικούς στόλου της Βόρειας Θάλασσας, το γεγονό ότι ζητούμε να μειωθούν κατά 30% οι καραβίδε στην περιοχή αυτή τη ε, Βόρειας Θάλασσας γύρω από την Ιρλανδία, αυτό θα καταστρέψει τον αλληλευτικό στόλο. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολλούς από εμά τα επιστημονικά αποτελέσματα δεν μας υποδεικνύουν μια τέτοια ανάγκη μείωσης των αλλιευμάτων. Η Βόρεια Ιρλανδία δεν χρειάζεται μία μείωση, χρειάζεται μία συνέχιση των αλλιευμάτων για του 2009 και το 2010 για τις καραβίδες στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η αληφτική δραστηριότητα στη Βόρεια Ιρλανδία. Θα σας δώσω και ένα από τα συμπεράσματα, ένα από τα αποτελέσματα μάλλον που θα συμβούν με τον τρόπο αυτό. Το κελκύλι είναι η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι στη Βόρεια Ιρλανδία με πληθυσμό περίπου 6.500 άτομα αυτή τη στιγμή. Κατά την περίοδο της οικονομικής κάμψης, όλες οι κύριες βιομηχανίες επλήγησαν ιδιαίτερα και η αλία είναι η τελευταία κύρια οικονομική δραστηριότητα που δίνει ακόμα θέσεις απασχόλησης. Μία μείωση κατά 30% λοιπόν στην αλλιευτική ικανότητα για τις γαρίδες του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι θα εξολοθρευτεί ο μικρός ακόμα αυτός στόλος που παραμένει στη Βόρεια Ιρλανδία. Εγώ μίλησα με τον αρμόδιο υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας για τα αλληλευτικά θέματα και ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον αρμόδιο υπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ιδιαίτερο αυτό θέμα. Είναι μια πραγματική κόκκινη γραμμή για την Βόρεια Ιλανδία και μια που δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε σε αυτό το στάδιο διαπραγματεύσεων. Ζητώ από την Κομισιόν να κοιτάξει και πάλι τα επιστημονικά στοιχεία και τις συνέπειες οι οποίες θα προωθούν από την πρότασή της. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας υποστηρίξω, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι για όλους από εμά τόσο σημαντικό, τόσο κεφαλαιόδες, που δεν μπορεί να διεκπαιρεωθεί σε δύο λεπτά, θα πρέπει να γίνει μια πραγματική και πλήρη συζήτηση. Ελπίζω ότι στην επόμενη φορά θα έχουμε χρόνο στη μέση διάταξη για να μπορέσουμε αντιστοίχω να το εξετάσουμε με αρκετό χρόνο. Ναι. Κυρία Ρότβιτς, είναι πρόθεσή μου να χρησιμοποιήσω το χρόνο που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εγώ το έθεσα στην μέση διάταξη γιατί μου φάνηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν το συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε πια συνεδριάσεις Επιτροπή Αλία μέχρι το Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα το Δεκέμβριο. Γι' αυτό υπήρχε το κατεπήγον να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη διεξοδικότητα, αλλά δεν ήταν δυνατό αυτό. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα να έχουμε μια ευρύτερη σημασία, σημασία συζήτηση σε κάποια στιγμή τη συνεδρίασή μα. Η Κομισιόν. Καταλαβαίνω το προβληματισμό σα. Όπω σα είπα, η διαχείριση τη αλληλεία πρέπει να δούμε τι κερδίζουμε βαχυπρόθεσμα και τι κερδίζουμε μακροπρόθεσμα. Ο, ο του Βορρά Όλος πέτυχε τους στόχους του. Είναι μες στα βιολογικά όρια. Ωραία, πολύ ωραία, ασφαλής. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να πάμε πέρα από τα αποθέματα, στο όριο της βιωσιμότητας, να πάμε πιο πέρα. Μεγίστε βιώσιμη απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλώνται καύσιμα, σπαταλώνται ανθρώπινη προσπάθεια, σπαταλάται κεφάλαιο η απόδοση μπορεί να είναι πιο μεγάλη και η αλληλεία να είναι πιο αποδοτική. Υπάρχουν ωφέλη αν κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η Κομισιό έκανε πρόταση για νοχυπρόθεσμη διαχείριση του γάδου της Βόρειας Θάλασσης, Χέιγκ, για μια αποτελεσματική αποδοτική χρήση των πόρων. Η πρόταση για τα ΤΑΚ που έχετε συμφωνεί απόλυτα με την πρότασή μας για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ναι, θα έχω μια απόλυτη βραχυπρόθεσμα. Ναι,